send once I had sent the email. That's lovely. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Καθίστε συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Χτες είχαμε μια εντατική συνεδρίαση και η σημερινή συνεδρίαση θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Υπήρξε μια φήμη ότι θα συνεδριάσουμε αύριο και την Πέμπτη, αλλά το διαψεύδω αυτό. Δεν θα υπάρξει συνεδρίαση της Επιτροπής μας ούτε αύριο ούτε την Πέμπτη πέραν τούτου. Θα δώσω το λόγο διακόπτει ο Dans eh Λοιπόν, προετοιμαστείτε να ακούσετε τον γενικό εισηγητή πρώτα, τον κύριο Γκάιερ, ο οποίος μετά από την συνεδρίαση κατά την οποία η κυρία Γεωργίευα παρουσίασε τις βασικές γραμμές για το 2017, ένας πολύ στενός προϋπολογισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε μάλιστα έξι εβδομάδες επιπλέον, αναβάλλοντας από τα μέσα Μαΐου στο τέλος Ιουνίου την παρουσίαση του σχεδίου της. Υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων την 4η Ιουλίου εν τω μεταξύ ο Γενικός Εισηγητής μας συνέταξε μια σύσταση η οποία συζητήθηκε χθε ε, σε μια πρώτη φάση με τους συντονιστές και σήμερα ο κύριος Γκάιερ θα μας παρουσιάσει αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες και θα μεταφέρει τις απόψεις του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε το λόγο, περιμένοντας λίγο, για να γεμίσουμε το χρόνο. Α, βλέπω να φτάνει μόλις ο κύριος Γκάιερ. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν την ουσία του σχεδίου σύστασης, το οποίο θα σταλεί στο Συμβούλιο, θα πιέσει θα έλεγα το Συμβούλιο και θα καταλάβει ότι το, το Συμβούλιο ελπίζουμε ότι οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δεν μπορεί να αγνοηθούν. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί λοιπόν αυτή η συζήτηση η οποία ξεκίνησε χθε ε, μεταξύ των συντονιστών. Ξέρετε και γνωρίζετε το σημείο της που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Κανονικά στην προηγούμενη Ολομέλεια θα έπρεπε να είχαμε ψηφίσει μια εντολή για τον τριμερή διάλογο οι οποίες συνεδριάσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα ε, την τρέχουσα εβδομάδα για να ανταλλάξουμε απόψεις με τα άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό. Η αναβολή του ευρωπαϊκού προπολογισμού τροποποίησε τη διαδικασία αυτή και τώρα θα κληθούμε να εφαρμόσουμε μια διαδικασία την οποία είχαμε εφαρμόσει και το 2014, όπου και υποπλήθηκε καθυστερημένα το σχέδιο προπολογισμού. Το Συμβούλιο άσκησε κάποιες πιέσεις ε, προκειμένου μάλλον ε, πιέστηκε να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και προκειμένου να ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο μαζί μας, ε, ο οποίος τριμερής διάλογος θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Έτσι, μάλλον φθινοπορεινός τριμερής διάλογος και όχι τόσο εαρινός. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε επί της εντολής αλλά ακολουθούμε τη διαδικασία του 2014 και θα αποστείλουμε ε, ένα letter of recommendation, μια επιστολή συστατική προς, τις, ε, προς τα άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού. Και φυσικά η επιστολή αυτή θα περιέχει και τα στοιχεία συμπληρωματικά της γνωμοδότησης των άλλων συναρμόδιων επιτροπών. Ε, Εμμανουέλ Φερνάντες ε, έθεσε χθε το θέμα του κατά πόσο θα μπορούσε αυτή η επιστολή να αναβαθμιστεί, να καταστεί έγγραφο εργασία, να έχει και μια θεσμική αξία και να αποτελεί και ένα σήμα κατά τη θέναν θέλετε του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια επιστολή στο όνομά μου, επί της οποίας έχουμε συμφωνήσει και με τους τονιστές χθες σε μια πρώτη συνάντηση. Αυτό το έγγραφτο, αυτή η επιστολή, δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερε πολιτικές καινοτομίες. δεδομένων και όσων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ως κατευθυντήριες γραμμές τον Μάρτιο. Άρα όλα τα σημεία τα οποία υπογραμμίστηκαν στην οδηγία αποτυπώνονται στην επιστολή από πολιτική αποψή. Φυσικά συμπληρώνονται και από τα αριθμητικά στοιχεία και τα όσα προβλέπει το σχέδιο προπολογισμού το 2017. Να σας υπενθυμίσω ότι στην οδηγία αποφασίσαμε ότι αναμένουμε οι δαπάνες για τους πρόσφυγες να μην μειωθούν. Αυτό και συνέβη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει στις τίτλους 3 και 4 και χρησιμοποιεί τα περιθώρια μέχρι τα ανατοτά όρια τα οποία προβλέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα εξαντλεί πλήρως και επιπλέον χρησιμοποιεί και επιπλέον μέσα, επιπλέον χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να συμπληρωθούν οι τίτλοι αυτοί. Επιπροσθέτως, υπάρχει έντονη κινητοποίηση και στον τίτλο 1α και αυτό αποτελεί προτεραιότητα του Κοινοβουλίου και φυσικά δεδομένης και της κρίσης της προσφυγικής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη στα μεγάλα πράγματα πρέπει να αποδείξει την αξία της και στα θέματα απασχόλησης για παράδειγμα, είναι απαραίτητη η κινητοποίηση του τίτλου 1α. Γενικά υπάρχει μια διαφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο για την προτεραιότητα των μέσων. Ποια θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, ποια όχι ιδιαίτερη. Αυτά δεν παίζουν ιδιαίτερη σημασία όμως στην συστατική μου επιστολή. Γιατί συμφωνούμε ότι η κινητοποίηση για την αγορά εργασίας, για την απασχόληση είναι απόλυτα απαραίτητη. Επίσης τονίζουμε ότι στον τίτλο 1β στην ε, πολιτική συνοχή ε, υπάρχει, υπάρχει και προβλέπεται σαφής μείωση των πληρωμών. Δεδομένης ε, και της κρίσης του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα πρέπει να μην προκαλέσουμε περαιτέρω προβλήματα, αλλά σίγουρα θα κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό δικαιολογείται και αιτιολογείται η στάση μας. Χθε λοιπόν στους συντονιστές ε, δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντιπαράθεση. Θα ήταν υπερβολικό να το πούμε αυτό. Υπάρχουν ωστόσο σε κάποια σημεία διαστάσεις απόψεων. για το πόσο ξεκάθαρο, για παράδειγμα, θα πρέπει να καταστεί τα πλαίσια του ΕΦΣΥ τα πράγματα δεδομένου ότι και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ΕΤΕΠ σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα της ε, χρηματοδότησης των ε, project, κατά πόσον τηρεί αυτή την αρχή της συμπληρωματικότητας. Ξεκίνησε λοιπόν μια συζήτηση για το ΕΦΣΥ. 8 δις ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εγγύηση του ΕΦΣΙ και από τα 8 δις αυτά έχουν κινητοποιηθεί μόνο 3,8 δις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε και να ε, εκχωρήσουμε, μάλλον να κινητοποιήσουμε πιο πολλά χρήματα για την χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ. Έχουμε και στο πλαίσιο αυτό το Connecting Europe Facility και τον ορίζοντα 2020. Και αυτά αποτελούν εύστοχα προγράμματα και μάλιστα προγράμματα τα οποία, μάλλον μέσα τα οποία α, κινούνται προς τη γενικότερη κατεύθυνση της υποστήριξης της αγοράς εργασίας. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά σε συνάρτηση και με το ΕΦΣΥ. Για να μην χρησιμοποιηθεί το ΕΦΣΥ δηλαδή στη θέση Επίσης, αναφέραμε πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα κατάσταση. Οι γενικές ανησυχίε σε ό,τι αφορά το σχέδιο προπολογισμού, εκφράστηκαν και επαναλαμβάνω επιγραμματικά μόνο τις γνωστές θέσεις. Μιλήσαμε για την κρίση στις πληρωμές. Αναφερθήκαμε στην κατάσταση που επικρατεί για τα οικονομικά μέσα, τα οποία εν μέρη δεν λειτουργούν όπως θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεκτρικό Συνέδριο. Το δείξαμε λοιπόν αυτό και εκφράσαμε μια ανησυχία για την ε, πιο εκτεταμένη χρήση των ε, δημοσιονομικών αυτών ε, μέτρων και το πόσο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτικό χαρακτήρα των μέσων αυτών και σε ό,τι αφορά τη χρήση επιδοτήσεων. Και έδειξαμε το θέμα το ότι πολλοί πολιτικοί τομεί ουσιαστικά δεν θα μπορούσαν να πετύχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα χωρίς τις ε, επιδοτήσεις και αυτοί πλήττονται πιο πολύ από κάθε, κάθε άλλο τομέα. Και δυστυχώς χθες αναγκάστηκα να φύγω και νωρίς, ε, γιατί ε, επισκέπτομαι, ξέρετε, όλες τις ε, συναρμόδιες επιτροπές και συζητώ με τους συναδέλφους ως ε, γενικό συζήτης και διοργανώσαμε λοιπόν μια συζήτηση, μια, μια κρόαση για τη μεταρρύθμιση της διαμορφώσεις του προϋπολογισμού και ξέρετε μου είναι οικία αυτά τα θέματα και θεωρώ ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, Επιστημόνων ξεκίνησαν λέγοντας ακριβώς αυτό το πράγμα. Αγαπητό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλετε το θέμα του προϋπολογισμού, αλλά η μετάβαση από επιδοτήσεις σε δημοσιονομικά εργαλεία είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι, για παράδειγμα, πολύ εξαρτώμενα από τις επιδοτήσεις ε, τα προγράμματα. Ενδεχομένως σε κάποιους τομείς να υπάρχουν και φατικές επιδράσεις. Πρόκειται και για μια άλλη μορφή οργάνωσης ε, του προϋπολογισμού. Και θεωρώ ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού καλά θα κάνει να εξετάσει και την ε, μόχλευση, την ικανότητα μόχλευσης, τον πρακτικό χαρακτήρα των μέσων αυτών, όχι μόνο από τεχνικής αυστηρά άποψης. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτεί, αλλά πρέπει βασικά να σκεφτεί η αρμόδια επιτροπή ότι πρόκειται για ένα εντελώ διαφορετικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του προπολογισμού και συνεπάγεται κάποια συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ε, μειονεκτήματα. Όταν μειώνει κανεί τι επιδοτήσει, ε, ε, γίνεται πολύ πιο ορισμένη η δυνατότητα επίτευξη κάποιων πολιτικών στόχων. Και αυτό πάντα παίζει ένα ρόλο. Α θυμηθούμε ιδιαίτερα ότι τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση του τελευταίου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου θέλησαν ε, να υποσκάψουν ε, τη σημασία της μείωσης των επιδοτήσεων προς την αρμόδια επιτροπή. Ουσιαστικά δηλαδή διατείνονταν ότι ναι μεν ε, θα μειωθεί το ποσό των επιδοτήσεων αλλά θα χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. και το φθινόπωρο θα συζητηθεί πάλι το μεσοπρόθεσμο το μεσονομικό πλαίσιο και συμφωνεί η Επιτροπή μα ότι προ το παρόν είναι καλή χρηματοδότηση του προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για το ερώτημα του κατά πόσον και πώ λειτουργούν αυτά τα χρήματα οικονομικά μέσα. Και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα πολιτικά, τις πολιτικά και τα, τους πολιτικούς και τους τεχνικούς προορισμούς που συνεπάγονται το σύστημα αυτό. Αυτό, εν συντομία, είναι το περιεχόμενο της επιστολής συστάσεων, το οποίο και συζητήσαμε με τους συναδέλφους χθε και φυσικά προσβλέπω και στα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισήγητα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θα πρέπει να γίνει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουμε πάρα πολύ ε, χρόνο. Ξέρετε ότι αργότερα θα υποδεχθούμε τον κύριο Μόντι. Βον, ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του και για την πρόταση που κάνει για τη σύσταση. Εγώ ήμουν υπεύθυνο για την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και ασχοληθήκαμε κυρίως με το 1β ανησυχώντας για τη μείωση 23% στο 1β, είναι πάρα πολύ μεγάλη η μείωση αυτή. Είναι σαφές ότι τα προγράμματα που καλύπτονται εδώ είναι μακροχρόνια προγράμματα, καθυστερεί η εκκίνησή τους, αλλά θα έχει προχωρήσει, θα έλεγα, το πρόγραμμα μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικές πιστώσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στην απαραίτητη ταχύτητα κροαζιέρας η οποία χρειάζεται. με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι θα το πετύχουμε και δεν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μείωση. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι βέβαιοι ότι τα ποσά αυτά θα καλύψουν τις δαπάνες ε, για τις πληρωμές του χρόνου. Δεν θα πρέπει κάθε φορά να πηγαίνουμε προς τα πίσω και δεν θέλω να επαληθευθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον προϋπολογισμό για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας τον επόμενο χρόνο. Yes, good morning. Thank you Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή για το έργο του, για την προσπάθειά του να έρθει αυτό το έγγραφο και το επικοδομητικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη συναντήση των σκιωδών εισηγητών με τον εισηγητή μας. Έχω κάποιες παρατηρήσεις για το έγγραφο αυτό και για τη θέση της ομάδας μου ως προς το σχέδιο προπολογισμού που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, ε, θα επεξεργαστούμε τον προπολογισμό του 2017 ταυτόχρονα με την αναθε... ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε ό,τι αποφαστεί στα πλαίσια της ενδιάμεση αναθεώρησης του ΠΔΠ θα πρέπει να εφαρμοστεί αμελητή και να συμπεριληφθεί αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του 2017. Και θα ήθελα να περιλάβουμε ρητή δήλωση για το σημείο αυτό στις συστάσεις του. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους κονδύλια, ε, συμφωνώ με τον κύριο Βόν. 23% ε, ήταν η μείωση στο 1β, στο κονδύλιο για τις ε, πιστώσεις πληρωμών. Λυπούμε για αυτή τη μείωση. Όταν μας παρουσίασε το σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολόγησε ότι δεν έχουμε άλλες πληρωμές από το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως είπε ο κύριος Βον, θα χρειαστούν κονδύλια από το χρόνο, γιατί τότε θα μπουν σε πριλή λειτουργία. Γι' αυτό και θέλουμε περισσότερε εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ την οποία απευθύνω έκκληση. Στη διοργανική συμφωνία που θα έχουμε για τι πληρωμέ στι αρχέ Σεπτεμβρίου, θα θέλαμε σαφή επιχειρήματα και εξηγήσει για το σημείο αυτό. Και επίση, δεν θα ήθελα και πάλι να συσσωρεύσουμε ανεξόφλητου λογαριασμού στα τέλη ε, του πολίτου δημοσιονομικού πλαίσιου του τρέχοντος όπως κάναμε πέρυσι. Επίσης θα πρέπει να μπορούμε να κινητοποιήσουμε το περιθώριο απρόβλεπτων αναγκών. Ε, σωστή ελαστικότητα που διεκδικήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας δίνει τον περιορισμό των ανώτατων ορίων του, της δημοσιονομικής γραμμής 3. Θα χρειαστεί κάποια παρα, παρέκταση των ανώτατων ορίων. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, μείνουμε στις προτεραιότητές μας, στην απασχόληση, στην καινοτομία, στην έρευνα Γι' αυτό και οι δημοσιονομικές γραμμές 1α και 1β είναι σημαντικές. Χαίρομαι που η συγκεκριτή συμπεριέλαβε στο έγγραφο μικρή αύξηση ε, στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σημαντικές αυξήσεις στις πιστώσεις πληρωμών για να στηρίξουμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Και οι αναφορές στην προσθετικότητα που έχουν τα κονδύλια του ΕΦΣΥ. Θα πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υποβληθεί φέτος το Σεπτέμβριο για να δημιουργήσουμε μια πιο σαφή εικόνα, γιατί ε, μέχρι στιγμή τα μόνα στοιχεία που είχαμε ήταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και φορούσαν το 2015. Αλλά μετά από ολιγόμενη μόνο λειτουργία του ΕΦΣΥ, θα πρέπει να δούμε αν είχε τι θετικό αντίκτυπο έχει στην οικονομία σε διαφορά αφορά τον όγκο των επενδύσεων και χρειαζόμαστε πιο ακριβείς αξιολογήσει για το επενδυτικό σχέδιο. Περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο. Επίση θα πρέπει να επαναφέρουμε τι περικοπές που έγιναν, να διορθώσουμε μάλλον τι περικοπέ που έγιναν στον ορίζοντα 2020 και στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε πολύ καλά σχόλια εκεί και ιδιαίτερα στον ορίζοντα 2020 εξαιτία τη έλλειψη πόρων δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Επίσης, για τις δημοσιονομικέ γραμμές 2 και 4, να προσέξουμε αυτό το θέμα του αποθεματικού πρόβλημα των αναγκών. Στο, στο κονδύλιο 2 για την γεωργία έχουμε αρκετό περιθώριο για να αντιμετωπίσουμε τη πιθανή κρίση στη γεωργία. Αλλιώ στα 3 και 4, στα κονδύλια, συμφωνούμε εν γέννη με τις παρατηρήσεις του εισηγητού. Το ανώτατο όριο του κονδυλίου 3 θα πρέπει να αυξηθεί. Επίσης ε, και στο, πάλι στο 3 θα πρέπει να βρούμε νέα κονδύλια. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ευχαριστώ κυρία Ιζαμπέλ Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική. Γιατί όντως για τη δημοσιονομική γραμμή 1β θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα κονδύλια της ε, συνοχής δεν είναι μόνο κονδύλια αλληλεγγύης, αλλά και πολύ σημαντικά επενδυτικά μέσα, γιατί αυτό φαίνεται να το ξεχνούμε από τότε που θεσπίστηκε το ΕΦΣΥ. Ξεχνούμε ότι και τα κονδύλια αυτά συμμετέχουν στις επενδύσεις, πολύ εξίσου αν όχι περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και η μείωση των πληρωμών και με τις καθυστερήσεις που έχουμε ήδη σημειώσει, ε, είναι ακατάλληλες για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ε, σε ό,τι αφορά το 2, το κονδύλιο 2, χρήση 50% του μισού δηλαδή περιθωρίου για την ΚΑΠ, Καλώς, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να βεβαιωθούμε ότι η κινητοποίηση αυτών των περιθωρίων απρόβλεπτων αναγκών για τη Γεωργία που αντιμετωπίζει διαδοχικές κρίσεις ε, να μην αποβεί τελικά εις βάρος των δικαιούχων των αποδεκτών. Ευχαριστώ κύριο Τονανό. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω στον ίδιο τόνο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τη μείωση το 23,5%. Ε, υπάρχουν προσδοκίες και πρόκειται για τη σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και των ε, τοπικών αρχών, το ε, Ταμείο Συνοχής. Πρέπει επιμείναμε προσφάτως ε, για τη χρήση ε, των ε, πιστώσεων τέτοιου είδους είναι η σχέση μεταξύ των τοπικών των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διακαθυστέρηση πληρωμών. Είναι μεγάλη η γραφειοκρατία πίσω από αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία που καθυστερεί τις πληρωμές αυτές και σήμερα Περί αυτού πρόκειται. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Πρέπει να υπάρξουν λύσεις ε, για την ε, απλοποίηση των διαδικασιών και για τους μηχανισμούς διασύνδεσης. Δεν είναι δυνατόν, ε, ακούσαμε χθε τους ερευνητές, έχουν προσδοκίες και είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνοδεύσει ε, την έρευνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεπρέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να υπενθυμίσω αυτό που είπα εχθές, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό για την κοινή γνώμη. Όλες ε, οι πιστώσεις για την κατηγορία 3 και για την κατηγορία 4 ε, θεωρούνται από κάποιους πολίτες ότι είναι υπέρ ε, ε, δράσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανυπεβεβαιώσουμε τις προτεραιότητές μας υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι στον τομέα αυτό πρέπει να έχουμε τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, υποστήριξη των επενδύσεων. Γι' αυτό ακριβώς εχθές είχαμε κάποιες διαφορές με τον φίλο συνεισηγητή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, βρούμε μία λύση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πέρα από το ΕΦΣΥ. Επίσης, το θέμα των νέων ε, πρέπει να είναι μία τεράστια προτεραιότητα του προϋπολογισμού του το Erasmus ε, Plus. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατηγορία 1α και ένα τμήμα του 1Β για μας είναι εξαιρετική σημασία. Προφανώς θα υπάρξουν τροπολογίες ε, τις οποίες θα υποβάλουν οι συνάδελφοι για την κατηγορία 2 γιατί είναι σαφές ότι στην κατηγορία 2 πρέπει να υπάρξει ένας χώρος που να επιτρέψει στους ε, γεωργούς ε, να βγουν από ε, την κρίση που προέκυψε από το εμπάργο της Ρωσίας, όπως της Ρωσίας και επίσης να καλύψουμε το πρόβλημα της παραγωγής γάλακτος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση για την βαρύτητα που θα έχουν οι πληρωμές. Τρία χρόνια ε, έχουμε διαπραγματεύσει στον τομέα του, ε, δημο, του προϋπολογισμού. Λες και ε, δεν είναι σημαντικό να είμαστε υπεύθυνοι για τις πληρωμές. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στις πληρωμές και συζητάμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να μας δημιουργεί πρόβλημα. Με έχει κουράσει ότι κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό των ε, πληρωμών για την ε, μείωση τώρα του 23,5% ε, ή πρόκειται για ε, μια οργάνωση σοβαρή η οποία έκανε σωστούς υπολογισμούς είτε όχι. Τίποτε δεν έγινε λοιπόν ε, για να γίνει καλύτερη διάρθρωση των πληρωμών για να μην βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου να έχουμε τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Εγώ δεν θα ήθελα να περάσω άλλη μια χρονιά να τσακώνομαι με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να τους λέμε δώστε μας λεφτά. Δεν είναι για μας τα λεφτά αυτά. Αυτό θέλω να, να είναι απολύτως σαφές εγώ δεν μιλάω πια για το θέμα των πληρωμών. Μιλάω για τις θετικές προτεραιότητες επί των οποίων πρέπει να επιτύχουμε αποτελέσματα. Και αν η Επιτροπή έκανε λάθος ε, στους υπολογισμούς της, πρέπει να κάνει σοβαρές ε, προτάσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης και εμείς να την υποστηρίξουμε κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση τη μονομερή και την οργάνωση τη μονομερή ε, των ε, ε, πληρωμών, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λάθος, πρέπει να το διορθώσει. Να σας υπενθυμίσω ότι μόνο μισή ώρα έχουμε ακόμη και έχουμε να καλύψουμε και τα υπόλοιπα τμήματα. Τέσσερις ακόμη θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ να είστε ε, σύντομοι. Ο κύριος Μονκά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή Γκάιερ ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν περισσότερα κονδύλια και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και να μεριμνήσουμε να είναι αποτελεσματικό το ΕΦΣΥ και να συμπληρώνει, να προστίθεται στα υπόλοιπα κοινοτικά κονδύλια και όχι να τα υποκαθιστά. Έχουμε κρίση και στις πληρωμές, ε, γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίση, να εξασφαλίσουμε πόρου για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και όχι από τραπεζικά δάνεια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει αρκετό διαθέσιμο κεφάλαιο και να μην αναζητούμε κονδύλια και χρηματοδότηση μόνο από τι κεφαλαίες Θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην ε, ε, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα τραπεζικά δάνεια. Επίσης, ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την Τραπεζική Ένωση που είναι απαραίτητη για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για τη μείωση των κινδύνων του τραπεζικού τομέα. Και να μην ε, ξεχνάμε και τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, γιατί αν θέλουμε σταθερό προπολογισμό, δεν μπορεί να μένουμε τόσο πίσω. Δεν μπορούμε να ειστερούμε τόσο πολύ στα θέματα αυτά. Εδώ και πολύ καιρό είχαμε τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους και κανονικά θα έπρεπε να, να πλησιάζουμε πια στο τέλος της. Φαίνεται όμως ότι μόνο στα τέλη του έτους θα έχουμε ε, περισσότερες πληροφορίες, αλλά δυστυχώς οι καθυστερήσεις αυτές είναι εις βάρος μας. Ο κύριος Φερνάντες. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Κατανοώ αυτά τα οποία είπε και ο Γεράρ Δεν πρέπει εμείς να θεωρήσουμε ότι μόνο οι πληρωμές είναι η προτεραιότητά μας, αλλά οι πολιτικές είναι η προτεραιότητά μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της. Έχουμε ζητήσει κάτι πολλές φορές και μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων θέλουμε ένα πρόγραμμα πληρωμών μέχρι το 2020 σε αυτή την πολυετή ε, προσπάθεια προγραμματισμού. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ξεχνάμε. Θέλουμε να υπευθυνοποιήσουμε λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στις πληρωμές. Ένας ερευνητής μας έλεγε χτες ότι περίμενε εδώ και ένα χρόνο ε, ε, μια πληρωμή, του έλειπε ένα έγγραφο και υποφελεί το από αυτό η Επιτροπή για να μην τον πληρώνει. Κυρία Νεριάντα, εγώ θα είμαι ακόμη πιο επιγραμματική γιατί συμφωνώ με του προλαλήσαντε για αυτά που είπαν ε, για την ε, ανεργία των νέων και να μην επικεντρωθούμε υπερβολικά στα μέτρα ασφάλειας. Συμφωνώ με τον κύριο Τεπρέ για το πρόβλημα που έχουμε στις πληρωμές, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν συνετό να μην αναλάβουμε κάποιες ευθύνες ε, αναφέροντας το σημείο αυτό, γιατί έτσι ίσως ε, επισκιάσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες και ιδιαίτερα τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Προσοχή να βρούμε τη σωστή ισορροπία και να μην παραμελήσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτή η πρότασή σα, απλώς να είμαστε συνετοί στην προσέγγιση και να, να δούμε τι θα γίνει με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο του 2020. Ελπίζω να ήμουν αρκετά επιγραμματική. Κύριος Μαραγκάλ, ευχαριστώ επιγραμματικά. Θεωρώ ότι το έγγραφο του κυρίου Γκέιερ είναι χρήσιμο γιατί μας βοηθάει να δούμε πώς αποστασιοποιηθήκαμε από την προηγούμενη μας θέση για την διάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και την πρώτη αυτή συγκεκριμενοποίηση μετά τις τελευταίες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια περισσότερο πολιτική παρά τεχνική συζήτηση. Προτεραιότητες, νέοι στόχοι, ε, δημοσιονομική ικανότητα για να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες ε, και απαιτήσει ε, που μας δημιούργησε η αδύρυτη πραγματικότητα. Και φυσικά προ... την αξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού, που ιδιαίτερα φέτος είναι πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε μπορούμε ως Κοινοβούλιο να διατρανώσουμε την ανησυχία μας και τις απαιτήσει μας να διορθωθούν, αλλά είναι προφανές ότι αυτό το θέμα αφορά δύο διαφορετικά και προσδιορισμένους κόσμους διαχείρισης. Πρώτον, τον κόσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεύτερον, τον κόσμο των κρατών μελών και την πραγματική του ικανότητα να διεκπαιρεώσουν ε, τα προγράμματα και τις δεσμεύσει που έχουν αναλάβει και ιδιαίτερα με τα κονδύλια του προπολογισμού. Επίση, ε, θα έπρεπε να συζητήσουμε και την ίδια έννοια τη σύλληψη του, της δημοσιονομικής διαχείρισης που βρίσκεται πίσω από αυτήν ακριβώς την ε, ανεπαρκή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, πολλές προκλήσεις και πιστεύω ότι αυτός ο προπολογισμό θα είναι ο πρώτος μετά την αναθεώρηση και όχι ο τελευταίος της προκαταρκτικής αναθεώρησης. Θα πρέπει να δούμε το εύση, το Έρασμος, τη νεολαία, ε, την, ε, τις κλιματικές αλλαγές, γιατί αυτό το ξεχάσαμε. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, απαιτήσει της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ό,τι αφορά το ποσοστό των δαπανών που θα πρέπει να αφιερώσουμε στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οπότε, και να, και να μην ξεχνούμε και την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια γιατί ζητήσαμε αυξήσει στο 1α, 1β, στου τομέ 3 και 4, υπέρβαση των ανώτατων ορίων. Θα είναι περίπλοκο αυτό και θα καθορίσει η συζήτηση το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εκατομμύρια πολίτε περιμένουν και θα πρέπει να δώσουμε λόγο σε αυτού. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριο Κιουλμέλ. Ε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Γιατί σε πάρα πολλά σημεία ε, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί του και είμαι βέβαιος ότι η ομάδα μου θα υποστηρίξει τα στοιχεία αυτά κατά συντριπτική πλειοψηφία. Ωστόσο, να τονίσω και το εξή. Δεν πιστεύω, όπω επεσήμαναν πολλοί, ότι πρόκειται για πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονό ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει μεγάλα ελλείμματα μεταξύ των δεσμεύσεων πληρωμών και των ε, μέσων πληρωμών τα οποία διατίθενται. Αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμεί ουσιαστικά είναι αυτοί που αποφασίζουμε τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μα απασχολεί εμά το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω και το εξή. Εννοείται ότι θεωρούμε ότι έχουμε δύο δυνατότητε να καλύψουμε το κενό αυτό. Αλλά δυστυχώ, εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα μιλάμε για την αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων. Έτσι θα μπορούσαμε να κλείσουμε το κενό αυτό. Άρα θα μπορούσαμε να κλείσουμε ε, και το κενό αυτό ε, μειώνοντα τι δεσμεύσει ε, και τις υποσχέσεις. Αυτό φυσικά φαίνεται ότι δεν είναι ευκταίο και επιθυμητό. Θα ήταν πάρα πολύ καλά φυσικά να τα είχαμε τα χρήματα αυτά, αλλά εφόσον τα είχαμε, αλλά αφού δεν τα έχουμε. Και μια και δεν έχουμε τα χρήματα για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις πληρωμές, μήπως θα έπρεπε να μειώσουμε τις δεσμεύσεις. Αυτό θα ήταν ευθύνη μας. Και άρα, τα πιο πολλά είναι σωστά από αυτά που λέει ο κύριος Γκάιερ, αλλά να μην ξεχνάμε τις αδρές γραμμές. Το έχει επαναλάβει αυτό ο κύριος Γκάιερ σε διάφορες περιστάσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις, ε, τα καθήκοντα που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να τα εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα, θα πρέπει να μας διαθέσουν τα, τους πόρους τα κρατημέλη. Ή τέλο, θα βρισκόμαστε ε, πάντα σε αυτό το σπαγκάτο, το οποίο δεν έχει διέξοδο. Ο κύριο Γκάιερ, εν συντομία. Πάρα πολύ σύντομα, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ όλους για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Χαίρομαι που ακούω ότι εντάξει μπορεί να έχουμε κάποιε διαφορέ ω προ τι λεπτομέρειε, αλλά γενικά η γενικότερη προσέγγιση μα βρίσκει σύμφωνο εδώ στο Κοινοβούλιο. Κινούμαστε προ την ίδια κατεύθυνση. Δεν έχω πολύ χρόνο στην ε, διάθεσή μου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να αναφέρω ένα μικρό στοιχείο, εν συντομία. Το οποίο και τονίζει αυτά που μόλι ανέφερε ο συνάδελφο Κολμέκ. Ανησυχώ, ανησυχώ. Κάπω γιατί θεωρώ ότι αν δεν ε, στείλουμε τώρα ένα σαφές μήνυμα για την ε, σύνδεση που υπάρχει μεταξύ την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και των ε, διαβολεύσεων που παίρνουν, που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι για την υπερβολική επιβάρυνση του προπολογισμού. Υπάρχει ευρεία σύμφωνια στα θεσμικά όργανα, ότι θα πρέπει να κάνουν πιο πολλά και να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα στον τομέα της κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Υπάρχουν και συμφωνία για το ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες αυτές ε, οι δραστηριότητε. Εκεί που επικρατεί διάσταση απόψεων είναι κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει με τους τρέχοντες πόρους, τους διαθέσιμους πόρους. ο κλάδος αυτός είναι υποχρηματοδοτούμενος και το μόνο που πρέπει να αποφύγουμε είναι να τον φορτώσουμε με επιπλέον καθήκοντα. Υπάρχει πολιτική ανάγκη να γίνει αυτό, δεν τον τη Αλλά ένα περαιτέρω πολιτικό ζήτημα στη συζήτηση είναι αυτό. Και όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και έχουν δίκιο, θεωρώ, τα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμών. Αν η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι, τα κράτη, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει πιο πολλά πράγματα στην τομέα τη ασφάλεια και τη ε, κοινή άμυνα, αυτό δεν γίνεται χωρί επιπλέον πόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν ε, ο δικός μου τομέας ευθύνης ε, να σας κάνω παρουσίαση για τα λοιπά τμήματα και όπως γνωρίζετε είναι τα 1, 2, 3, 4 και 7 1,4 δις ευρώ τίποτε σπουδαίο δηλαδή θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά μικρότερη σημασία προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε κατά την διαδικασία που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την ΟΚΕ. αυτό έχει κάποια επίδραση και στο δικό μας προϋπολογισμό, γιατί μειώθηκε κάπως ο προϋπολογισμός ο δικός μας ε, και αυτό έχει μία έμεση επίδραση, έναν έμεσο αντίκτυπο στο δικό μας προϋπολογισμό και είναι σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι όταν θα ε, παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός, ε, ίσως καλύτερα με ανταλλαγή επιστολών αντί για την κανονική δημοσιονομική διαδικασία. Δεύτερον, όταν μιλούμε για το ελεγκτικό συνέδριο, συγγνώμη, για το δικαστήριο, νομίζω ότι είναι, περισσό, είναι πιο σημαντικό να υπάρξουν περισσότερες θέσεις ε, μετάφρασης ε, αντί να γίνεται εξωτερική ανάθεση ε, πολύ περίπλοκων νομικών κειμένων και βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές σε σχέση με αυτό στα διάφορα όργανα. Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται από τους υπαλλήλους μεταφραστές, σε, άλλους, σε άλλες περιπτώσεις κάνουμε εξωτερική ανάθεση των κειμένων αυτών. Εν πάση περιπτώσει, είμαι Βέβαιος ότι θα βρεθούν ε, οι απαραίτητες λύσεις ε, κατά τις ε, επερχόμενες συζητήσεις και με χαρά θα περιμένω, με αγωνία θα περιμένω τις προτάσεις των συναδέλφων για όσα θα συμβούν την επόμενη χρονιά. Κύριε Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συμφωνώ με τα συμπεράσματά του. Δύο ακόμη σχόλια. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε μειώσει κατά 5% ε, περίπου ε, το προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό ε, γιατί μειώνεται συχνά ε, το προσωπικό, ειδικά στο δικαστήριο και γίνονται ε, εξωτερικές αναθέσεις συνεχώς κάτι το οποίο μειώνει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών οργάνων. Πρέπει να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, είτε ή να ακολουθήσουμε τον τρόπο τον κανονικό, την κανονική διαδικασία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει την άποψη ότι θα γίνουν μεταφορές πιστώσεων. Πέρσι είπαμε ότι ο δείκτης θα ήταν μικρότερος από αυτόν που αναμέναμε και σήμερα λέμε ότι ο τιμάριθμος έχει όντως ε, υπερεκτιμηθεί. Πώς ε, θα καταφέρουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, αξιοπιστία μας. Ο κύριος Δενανό, σύντομα. Ναι, κοιτάξτε, ε, και εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις δύο παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Τάραντ. Και ο κύριος Μάνκα μόλις είπε αυτό που ήθελα να πω για την μη εξωτερική ανάθεση των διερμηνέων. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα της ΟΚΕ, Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και ξέρω τι σημασία έχει για τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις τοπικές αρχές αυτό το όργανο και καταλαβαίνω τις δικές τους προσδοκίες. Πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφωνώ με την άποψη του κυρίου ε, Τάραντ σε σχέση με την ε, ε, σημασία που πρέπει να δώσουμε στη μείωση των πιστώσεων αυτών. Μία ακόμη φορά λοιπόν επικροτώ την εξαιρετική δουλειά ε, των εισηγητών μας, του κυρίου Τάραντ και του κυρίου ε, Γκάγερ. Να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση. Θα έχετε δύσκολο έργο απέναντι στο Συμβούλιο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε μας κάνουν να σκεφτούν ε, ότι το Συμβούλιο θα μειώσει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών. Πολύ έντονη πίεση λοιπόν, κύριε Γκέιερ, θα πρέπει να ασκήσετε κατά τις συστάσεις. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα Φερνάντε Γκάιερ για τι ε, προπαρασκευαστικέ δράσει και τα πιλωτικά προγράμματα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σύντομοι, ε, κύριοι εισηγητέ, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά ακόμη. Έχουμε τον αριθμό των, ε, προγραμμάτων για το, των πιλωτικών προγραμμάτων για το 2017, αλλά δεν έχουμε την αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα την έχουμε το Σεπτέμβρη μόνο. Μέσα Ιουλίου θα γνωρίζουμε. Μέσα Ιουλίου. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ για να λάβουμε γνώση. Κύριε Φερνάντες. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι ε, τηλεγραφικός μετά το, τη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2017 του κ. Γκάιερ και τα πολιτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικέ δράσει είναι σημαντικά ζητήματα για την προετοιμασία των νέων πολιτικών και για τη δυνατότητα που έχουμε να ε, προτείνουμε λύσεις που στη συνέχεια θα μεταφραστούν σε προγράμματα. Όλα, έχουν, όλα έχουν ξεκινήσει και όλα τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με τα απαραίτητα μέσα και πόρους για να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Για το 2017 και με τα περιθώρια που έχουμε είναι σίγουρο ότι και εγώ θα προσπαθήσω να πετύχουμε μια καλύτερη κατανομή και να δώσουμε προτεραιότητα στις, στα καλύτερα προγράμματα. Φροντίζοντας όσο περισσότερα ποιοτικά πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικές δράσεις να χρηματοδοτηθούν. Έτσι θα παρουσιάσουμε τις ιδέες μας και θα τις μεταφράσουμε σε προγράμματα δείχνοντας τους ε, πολίτες και αναμειγνύοντας τους ε, ακόμη με δείχνοντας λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να αποβεί χρήσιμη και να εξυπηρετεί τους πολίτες της. Ευχαριστώ κύριος Γκάιερ. Νομίζω ότι και εγώ θα μπορούσα να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση, όπως και ο προλαλής σας. Μανουέλ Φερνάντες, έχουμε 321 νέε προτάσει. Και αν ρίξουμε μια ματιά στις αναλήψει υποχρεώσεων, θα απαιτούσαν 487 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότησή του. Δύσκολο εγχείρημα με τον τωρινό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιοριστούμε λοιπόν στα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, ε, κάνοντας μία εράρχηση και εστιάζοντας τα πιο σημαντικά. Ανάλογα και με την αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επόμενη εβδομάδα ίσως κάνουμε πιο σχολαστική ανάλυση και θα επωφεληθούμε και από τις θερινές διακοπές ε, για να καταστελάξουμε σε ορισμένα θέματα. Επίσης, θα ήθελα να επιμείνω σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα στοιχήσει 25 εκατομμύρια και η ερώτηση που θα σας θέσω είναι περισσότερο ρητορική για το αν αξίζει τον κόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Σίγουρα αξίζει και με τον μικρό προϋπολογισμό που έχουμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα. Άλλωστε έχουμε 80 εκατομμύρια που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείνει σε αυτά τα 25 εκατομμύρια για την έρευνα στα θέματα της άμυνας, αυτά θα πρέπει να εκπίπτουν από τη σύνηθις ποσοστός για τη χρηματοδότηση των πιλωτικών προγραμμάτων για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Αυτά τα 25 εκατομμύρια για την άμυνα θα πρέπει να είναι ξεχωριστά. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα υπόλοιπα πιλωτικά προγράμματα, γιατί και τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις είναι οι μικροί μοχλοί που έχουν απομείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δείξει ότι έχει πραγματικά μια προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει. Ο κύριος Δεπρέ. Θα είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο εισηγητή μας. Ο αριθμός των προπαρασκευαστικών δράσεων που προτείνεται αποδεικνύει την κοινοβουλευτική εφάνταστη δραστηριότητά μας. Βλέπω ότι έχουν υπάρξει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο 43 προτάσεις. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι τα 25 εκατομμύρια που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν τμήμα των πιλωτικών προγραμμάτων το βάφτισαν πιλωτικό πρόγραμμα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει εκεί. Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν λοιπόν τα 25 εκατομμύρια. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια επιλογή που έχουμε μπροστά μας, να χρησιμοποιήσουμε με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής κάποια επιπλέον κριτήρια. Δηλαδή, θα ε, δεχθούμε αυτά τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως τα καλύτερα. Και αν τυχόν επιλέξουμε και άλλα, τότε πρέπει να το τεκμηριώσουμε. Έτσι κι αλλιώ θα είναι δύσκολο εμείς ε, να δεχθούμε τα προγράμματα που έχουν χαρακτηριστεί πρώτου επίπεδου, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα. Διαρωτώ λοιπόν τι διαδικασία θα ακολουθήσουμε γιατί αλλιώς θα λειτουργήσουμε λίγο αυθαίρετα. Ο πρόεδρος λέει ότι ίσως θα πρέπει να επαληθεύσουμε και τη συμβατότητα με τους κυρίαρχους στόχους που έχουμε θέσει του κάθε προγράμματος. Πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα σαφής ανάμεσα στις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στις συστάσεις του Γενικού Εισηγητή μας, μεταφέρει τις απόψεις των πολιτικών ομάδων και αυτός να είναι ένας από τους παράγοντες επιλογής Συμβατότητα δηλαδή με τους ε, κυρίαρχους στόχους. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, θα σταθούμε εδώ, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τώρα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Χριστοφόρου για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με την αξιολόγηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επισημάνω κύριε Πρόεδρε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ταμείο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε το 2002 για αντιμετώπιση των καταστροφών και έκτοτε αντιμετωπίστηκαν μέσω του Ταμείου 69 καταστροφές σε 24 χώρες και παραχωρήθησαν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2014 και με πρωτοβουλία της δικής μας Επιτροπής αναθεωρήθηκαν οι κανονισμοί, απλοποιήθηκαν και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες. Δύο σημαντικές βελτιώσεις που είχε το Ταμείο είναι ότι με πρωτοβουλία της Επιτροπής δική μας πρωτοβουλία ε, παραχωρούνται προκαταβολές 10% στην εκτιμόμενη καταστροφή που έγινε σε μια χώρα μέλος για να υπάρχει δυνατότητα άμεση ανταπόκριση στις ζημίες. Όμως, και το αναφέρουμε μέσα στην γνωμοδότηση, παραμένει τεράστιος χρόνος από την ολική διευθέτηση του όλου ζητήματος και απαιτούμε όπως απλοποιηθούν οι διαδικασίες στα διάφορα στάδια για να μπορεί να αποδίδεται άμεσα η αποζημίωση στι διάφορες καταστροφές. Επίση υπήρχε ένα πρόβλημα με τι περιφερειακέ καταστροφέ. Εκεί όσε αιτήσει υποβλήθηκαν απερίφθησαν εξαιτία του ότι δεν μπορούν να πληρούν τα κριτήρια οι περιφερειακέ καταστροφέ. Τώρα το μόνο κριτήριο που έμεινε είναι αυτέ οι περιφερειακέ καταστροφέ στην περιφέρεια που γίνονται να είναι μόνο το 1,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο ω το σύλλη για να μπορέσει να αποζημιωθεί αυτή η περιοχή και υπήρξαν αιτήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι παραμένει ακόμα ένα πρόβλημα για να μπορέσει μια χώρα να χρηματοδοτηθεί, ιδιαίτερα οι μικρέ χώρε, πρέπει η καταστροφή να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αναφέρω ένα παράδειγμα πρόσφατα και για τη χώρα μου. Υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές που ανέρχονται σε 40-50 εκατομμύρια. Όμως για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μια χώρα μικρή όπως η Κύπρος πρέπει να είναι τουλάχιστον η καταστροφή πάνω από 100 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ευελιξία είτε η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά, είτε να αλλάξουμε αυτόν τον όριο που τίθεται και αποκλεί πολλέ χώρε, δηλαδή να μην φτάνουμε στο σημείο να παρακαλούμε να είναι μεγάλε οι καταστροφέ για να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Αν είναι μικρέ οι καταστροφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Υπάρχουν παρατηρήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφό μας τον κύριο Χριστοφόρου για την παρουσίαση που μας έκανε και τις πολύ ε, φρόνιμες συνετές παρατηρήσεις. Είναι κάπως αυθαίρετο το ελάχιστο αυτό όριο που είναι κυρίως σε μια ενθάρρυνση. Θα πρέπει κανείς να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια για να έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοια συζήτηση και να είναι όλα θέμα ποσοστού. Δεν βλέπω κανένα να ζητά το λόγο, κάτι που αποδεικνύει ότι ο εισηγητής κάλυψε απόλυτα τους συναδέλφους και εξέφρασε το κοινό αίσθημα. Η προθεσμία λήγει αύριο το μεσημέρι για τις τροπολογίες. Την 1η Σεπτεμβρίου θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση και θα ψηφίσουμε. Στις 8 Σεπτεμβρίου η αρμόδια κατουσία Επιτροπή Ρέγγι θα ψηφίσει τη δική της έκθεση και θα περάσει στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου η σχετική έκθεση. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, τις πιθανές εξελίξεις και τις προσαρμογές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτης γνωμαδότης είναι ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάνδες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κρίναμε σκόπιμο ε, αμέσως μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, να προχωρήσουμε και ήδη από τον Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθούμε επί τριών γνωμοδοτήσεων που είναι ένα πακέτο. Η έκθεση Μπερές Μπέγκε που συζητήσαμε χθε και θα ξανασυζητήσουμε αργότερα από τις 11.30 μέχρι τις 1. Έχουμε την έκθεση Μπροκ Μπρέσο, BB έκθεση και επίσης και την τρίτη έκθεση, τμήμα του πακέτου, την έκθεση Verhofstadt. Αυτές οι τρεις εκθέσεις κατά πάσα πιθανότητα θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι συμβατοί προσανατολισμοί των τριών εκθέσεων και να συστήσουν την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και ίσως και να πρωτοστατήσει στη συζήτηση για τη διακυβέρνηση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Μάλιστα το Eurogroup για πρώτη φορά ε, θα επιβάλλει κυρώσεις δείχνοντας το κύρος του. Και αν κρίνουμε από τις ε, σημερινές δηλώσεις του Επιτρόπου, <laughs> το ποσοστό των ε, κυρώσεων θα είναι 0%. Μηδενικό το ποσοστό του προστίμου. Δεν είναι αξιοσημείωτο. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να κάνω το ερώτημα, να θέσω το ερώτημα ποια είναι τα κράτη-μέλη που ήταν ε, οι πρώτες που δεν σεβάστηκαν ε, τους κανόνες, η Γαλλία, η Γερμανία και καμία απολύτως κύρωση. Κύρωση μηδενική, όπως είπατε. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και μία φράση ε, κάποιος πάρα πολύ σημαντικός στην Ήπειρο ότι η Γαλλία δεν έχει κυρώσει γιατί είναι η Γαλλία. Και αν ε, ε, ακολουθήσουμε την αρχή της ισότητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε χώρα, κάθε χώρα ε, δεν έχει ε, δικαίωμα, δεν, δεν πρέπει να υποστεί κυρώσεις, ε, διακόπτει ο Πρόεδρος, για να επαναλάβω αυτό που είπα εχθές το βράδυ. Έχουμε έναν κανονισμό συνειδιοκτησίας του ευρώ ε, του οποίου ηγήθηκαν η Γαλλία και η Γερμανία. Δεν υπήρξαν ποτέ κυρώσεις. Τώρα όμως αλλάζει τα πράγματα. Τώρα έχουμε κυρώσεις, αλλά κυρώσεις με ε, μηδενικό ποσοστό. Είναι κάτι το οποίο ίσως ε, σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κυβέρνηση της Ευρωζώνης. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Φερνάντες, εγώ Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το συμπέρασμα με τον τρόπο που το καταλαβαίνει ο Πρόεδρος και θα ήθελα να περάσω στο δικό μου το θέμα. Αλλά θα ήταν μια συζήτηση αυτό που αναφέρατε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί ακόμη μια, και μια μηδενική ε, κύρωση είναι μια κύρωση και θα μπορούσε να είχε αρνητικές συνέπειες. Δεν θα μπω ε, στις λεπτομέρειες ε, αυτού του ζητήματος, γιατί θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Πορτογαλία-Γαλλία όμως ένα μηδέν ήταν το αποτέλεσμα. Ναι, ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήμουν και στο γήπεδο όταν έγινε ένα μηδέν που αξίζαμε πραγματικά. Να μην κάνουμε ούτε αυτή τη συζήτηση όμως. Λοιπόν, θα μιλήσω τώρα πορτογαλικά. Το χρονοδιάγραμμα επισπεύστηκε. Αρχικά προβλεπόταν για τον Οκτώβριο η παρουσίαση της δικής μας θέσης και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέρφους. Βέβαια, οι περισσότεροι πήγαν στις συνεδριάσεις που έχουν ψηφοφορίες. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους ε, να συμβάλλουμε τις παρατηρήσεις τους ε, στην έκθεση, στην γνωμοδότηση. Ε, αυτό που προτείνω είναι απλό. Να διατηρήσουμε τις, ε, οι προκλήσεις διατηρούνται, για να μην πω ότι αυξήθηκαν. Παγκοσμιοποίηση, κλιματικές αλλαγές, δημογραφικό πρόβλημα, ενεργειακή εξάρτηση, ανεπάρκεια των φυσικών πόρων. Όλες αυτές οι προκλήσεις ε, εξακολουθούν να ισχύουν. Και οι στόχοι μας παραμένουν για την παιδεία, για την απασχόληση, την καινοτομία, την έρευνα, την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, το μητριασμού των κλιματικών αλλαγών. Εξακολουθούν να ισχύουν όλοι αυτοί οι στόχοι. Η στρατηγική του 2020 δεν θα τερματιστεί το 2020, θα συνεχιστεί και πέρα από τον χρονικό αυτό ορίζοντα. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις ε, και να έχουμε ευφύ, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Και για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας θα πρέπει να εφοδιαστούμε με τα απαραίτητα μέσα. Και εδώ είναι το πρώτο βασικό σημείο. Οι διαστάσει στο μέγεθος του προϋπολογισμού. 1% του καθάριστο χώριο προϊόντος για τον ενωσιακό προϋπολογισμό δεν αρκεί για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ένα άλλο σημείο αφορά την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ του ενωσιακού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών για να δημιουργήσουμε συνέργειες και να καταφέρουμε και πάλι να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ένα συναφές θέμα αφορά την ανυπάρκεια των δημοσιονομικών πόρων. Είναι πενιχρός ο προϋπολογισμός. Χρειαζόμαστε και πραγματικούς ίδιους πόρους. Και αυτό δεν το επιβάλλω μόνο οι συνθήκες, αλλά η πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περιμένουμε και τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό. Και η υπευθυνότητα είναι σημαντικό ζήτημα επίσης, η ευθύνη. Στο μέτρο που τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν δεσμεύσεις δεν θα πρέπει να μένουν αυτές τα χαρτιά. Θα πρέπει να τηρούνται, να μην αθετούνται υποχρεώσεις και υποσχέσεις. Σεβασμός των υποχρεώσεων προποθέτει σεβασμό και του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και έχουμε και το θέμα του 5% και το ζήτημα της ευελιξίας. Οι, οι πόροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και που έχουν απελευθερωθεί δεν θα πρέπει να χάνονται, να πάνε χαμένα αυτά τα κονδύλια που δεν έχουμε αξιοποιήσει, που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά να μεταφέρονται στον προπολογισμό του επόμενου έτους. Βέβαια θέλουμε οι αναλήψεις υποχρεώσεων να τηρούνται κατά 100%. Αλλά και οι πληρωμές να γίνονται πλήρως. Να δηλαδή στο 100% και η αναλήψη υποχρεώσεων και οι πληρωμές. Επίσης, έκτακτες καταστάσεις, σε απρόβλεπτες καταστάσεις θα πρέπει ε, να προβλέπουμε έκτακτους πόρους και να υπάρχει δυνατότητα υπέρβαση των ανώτατων ορίων του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, εφόσον πρόκειται για έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. Και επίσης τα ειδικά μέσα που έχουμε θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιλαμβανόμαστε και να έχουμε κοινή ερμηνεία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εκεί διαφωνούμε, από το Συμβούλιο, με, διαφωνούμε με το Συμβούλιο για αυτά τα ειδικά μέσα και κατά πόσο είναι εκτός του, των ορίων. Γιατί αν ήταν να συμπεριλαμβάνονται στα, στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν θα είχαν αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα. Από τη στιγμή που είναι ειδικά μέσα, εξορισμού εκπίπτουν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό δεν το καταλαβαίνει το Συμβούλιο. Επίσης, όλο το δημοσιονομικό πλεόνασμα ενός έτους θα πρέπει να μεταφέρεται, επαναλαμβάνω, στο επόμενο έτος. Ένα άλλο θέμα που ανέκαθεν διεκδικούσαμε ήταν η ενότητα του προϋπολογισμού και η εφαρμογή της κοινοτική μεθόδου. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να δίνουμε προβάδισμα στα trust funds, σε αμοιβά κεφάλαια και σε ad hoc μηχανισμούς εκτός του προϋπολογισμού, χωρίς συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χωρίς εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένας ίσως τρόπος για να ξεπερνάμε το 1% του ΑΕΧ. Γιατί για τα κράτη-μέλη είναι το 1% για να ξεπεράσουμε το 1% χρησιμοποιούμε τη διακυβερνητική μέθοδο. Και ξεφεύγουμε από τον προπολογισμό, αλλά έχουμε ιδιαίτερους κανόνες. Ο μηχανισμός για την ενίσχυση των προσφύγων στην Τουρκία ε, ε, και οι συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτόν δεν συνυπολογίζονται στο έλλειμμα. Αν όμως τα κράτη-μέλη θέλουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες μέσω του προϋπολογισμού, αυτό το κονδύλιο που θα αφιερώσουν συνυπολογίζεται στο έλλειμμά τους. Άρα έχουμε διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με το κατά πόσο το μέσο, τα, τα, μέσα, οι μηχανισμοί εμπίπτουν ή εκπίπτουν από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ισχύουν κάποιες ε, εξαιρέσεις μέσω της διακυβερνητικής μεθόδου χωρίς να γίνεται σεβαστή η κοινοτική μέθοδος. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό που, για τον προϋπολογισμό είναι η απλότητα και η διαφάνεια. Και όταν μιλούμε για απλό και διαφανή προϋπολογισμό θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να είναι γνωστό πώς χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός και αυτό ισχύει για όλες τις αποζημιώσεις. Δεν έχει νόημα ένα κράτος να έχει μια εισφορά και να λαμβάνει μετά μια επιταγή 66% της εισφοράς του. Γιατί τελικά αυτό που ακούγεται δεν είναι η διαφορά αλλά το σύνολο. Και αυτοί που θέλουν να καταπολεμήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν το 100% με το 66%. Δεν μιλούν για την καθαρή συνεισφορά. και δεν μιλούν ε, για την επιστροφή. Απλώς ε, αναφέρονται στο αρχικό ποσό. Όλα αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και αυτά επισημένω στην γνωμοδότησή μου. Αυτές είναι οι προκατακτικές μου σκέψεις και περιμένω και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα έπρεπε τόσο γρήγορα να συντάξω την γνωμοδότηση, αλλά επαναλαμβάνω, επισπεύστηκε η διαδικασία εξαιτία των τελευταίων εξελίξεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πατρίσια Σουλίν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Φερνάντες για την παρουσίαση της γνωμοδότησης, για την γνωμοδότηση αυτή τις προσαρμογές στο θεσμικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις, όχι μόνο λόγω της μετανάστευσης. Νομίζω ότι είναι κάπως ανησυχητικά αυτά που συμβαίνουν στον τομέα της ε, ανεργίας των νέων. περίπου 7 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι, σύμφωνα με τα τελευταία ε, δεδομένα. Συζητάμε το θέμα ε, των ιδίων πόρων εδώ και μεγάλο χρονικό ε, διάστημα. Δεν έχουμε ακόμη λύσει το πρόβλημα αυτό. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα ε, συναντήσουμε σε λίγο τον Μάριο Μόντι που είναι ο επικεφαλής της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό και πραγματικά αναμένω με αγωνία τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι οι δημοσιονομικές ανησυχίες έχουν ε, άμεση σχέση και με το θέμα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στα επόμενα δύο χρόνια και επειδή πληρώνει περίπου 5 δις ε, ευρώ στον ε, προϋπολογισμό της Ένωσης, αυτό δημιουργεί ερωτήματα. Πώς θα προετοιμαστούμε για την κατάσταση αυτή. Έχουμε προβλέψει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ε, θα μειωθούν κάποια ποσά για κάποια προγράμματα ή αυτά τα 5 δισεκατομμύρια θα αντισταθμιστούν από τη χρήση μιας κλίδας κατανομής των κρατών μελών που θα πληρώσουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Βέβαια, αυτή δεν είναι η μόνη δυνατή λύση αν η κλίδα ε, κατανομής δεν επιβεβαιωθεί σε επίπεδο ένωσης, νομίζω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να συζητηθεί ευθύς αμέσως παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο συνήθως αναφέρεται στο πλαίσιο άλλου χρονοδιαγράμματος 2016-2017. Πρέπει να αντιδράσουμε σύντομα. Έτερη μου ανησυχία έχει να κάνει με τους οικονομικούς δείκτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι οποίοι παρουσιάζουν φθήνουσα πορεία και νομίζω ότι αυτό θα μειώσει και τους εθνικούς προϋπολογισμούς κατά συνέπεια. Αυτό θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να πληρώσουν λιγότερα στον ευρωπαϊκό, προϋπολογισμό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Σε κάθε οικονομική κρίση πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ε, διαφθοράς, ε, της φόροδιαφυγής ε, και Επίσης με απασχολεί το κατά πόσο είναι κατάλληλα, κατάλληλες οι διάφορες πολιτικές και τα διάφορα προγράμματα ε, και το κατά πόσο ο αντίκτυπος ε, σε αυτά έχει υπολογιστεί. Ελπίζω να μην ακούγομαι πολύ ε, απεσιόδοξη, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα προβλήματα που θα έχουμε να λύσουμε στο μέλλον. Κύριος Δενανό, ευχαριστώ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την έκθεση του κυρίου ε, Φερνάντες. Δύο, τρία ζητήματα μου φαίνονται πολύ σημαντικά. Πρώτον, το θέμα της μεταφοράς ε, των ε, πλεονασμάτων. Νομίζω ότι είναι η μοναδική περίπτωση που επιστρέφουν τα χρήματα στη τσέπη του φορολογούμενου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, σημεία σύγκλησης και η κατάσταση, η, η κατεπίγουσες περιπτώσεις. Ε, η απασχόληση των νέων για μένα είναι κάτι το κατεπίγον. Επίσης, η δημοσιονομική ε, ενότητα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απολύτως ε, ως προς αυτά, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα αυτής της συνειδιοκτησίας του ευρώ που αναφέρθηκε προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι μια συνειδιοκτησία στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε έργα όμως, ούτε ένα βαψιματάκι, ένα μερεμέτι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια πλήρη ανακαίνιση γι' αυτό συμφωνώ απολύτως με την ε, εκβάθρον ε, ανανέωση της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κολμέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρήσω, μάλλον να συγχαρώ τον συνάδελφο που κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αντίθετα με το ποδόσφαιρο, όπου συνήθως ε, μετά τη λήξη ενός ε, μάτς ε, αυτό που μένει είναι μόνο το αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα ξεχνιούνται. Ε, από πολιτικής άποψης ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά για όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση και μετά η ζωή συνεχίζεται και δεν έγινε τίποτα. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε το πώς επηρεάζει αυτά τα πράγματα. Και όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ εύστοχα κύριε Πρόεδρε, όταν υπάρχουν ρυθμίσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ε, όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις και μάλιστα επί μακρόν, επανειλημμένα απειλείται το συνολικό οικοδομήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν η δικαιολογία είναι ότι κάποτε κάποια στιγμή έγινε ένα σφάλμα και γι' αυτό διαιωνίζεται η διάπραξη τέτοιων σφαλμάτων είναι ουσιαστικά σαν να είναι κάπου τυπωμένες οι συνθήκες αλλά να μην υπάρχουν, να μην υφίστανται και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν μιλώντας για την ε, θεσμική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμού να λάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη, ναι. προκειμένου να είναι όλες οι διαστάσεις αυτές διαφανείς και αυτό δεν ισχύει σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Μόνο λίγοι εμπειρογνώμονες κατανοούν τα θέματα προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπόλοιποι είναι σε βαθύ σκοτάδι αναφέρθηκε για το θέμα της, ε, των καθαρών και μεικτών εισφορών. Αυτό ε, πολλοί δεν το κατανοούν. Δεν αφαιρείται από το ακαθάριστο, το καθαρό ε, ποσό και μετά καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Και θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής. Μήπως στην περίσταση αυτή δεν θα πρέπει να επιδείξουμε τόλμη και θάρρος, προκειμένου από κοινού να κάτσουμε, να σκεφτούμε το πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε δομικά, αντριφαντικά θέματα από πλευρά προπολογισμού. Έχει νόημα, για παράδειγμα, η Γερμανία που είναι ο μεγαλύτερο εισφορέα. Ε, και ομολογώ ότι η Γερμανία α, είναι ο μεγαλύτερος εισφορέας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν κάθε χρόνο δίνουμε 30 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε 14-16 δισεκατομμύρια α, ως αντίκρισμα, μήπως θα πρέπει να δίνουμε λιγότερα για να είναι πιο σαφής και πιο διαφανής ο προϋπολογισμός, να είναι πιο απλά τα πράγματα και να είναι σαφές το ποιος χρηματοδοτεί τι. Το θέμα δεν είναι προς Θεού να περιοριστούν οι εισφορές, γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εισφορές αυτές, αλλά χρειάζεται μια απλοποίηση και δεν καταλαβαίνω γιατί ένας αγρότης στο Μαλένα Δρυμό λαμβάνει μια επιδότηση η οποία περνάει από έναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί κάλλιστα από το εθνικό ή το ομοσπονδιακό, από το ομοσπονδιακό ή το ομοσπονδιακό επίπεδο. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει, να μια απίσχναση και απλοποίηση του προπολογισμού. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Δεν βλέπω να κάνει άλλο το λόγο για το θέμα του, του προπολογισμού και τη ενότητα του προπολογισμού. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάστηκε ένας πίνακας ο οποίο είχε προετοιμαστεί από τη γραμματεία και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το πράγμα. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Με όλα αυτά τα ειδικά μέσα, με τα επιμέρους ταμεία εγγυήσεων, με τους μηχανισμούς χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, με τα trust funds, με τα διάφορα facilities, ε, γενικά έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Νομίζω ότι βασικός κανόνας σε μια δημοκρατία είναι οι πολίτες να είναι σε θέση να κατανοήσουν το τι είναι ο προϋπολογισμός, ώστε οφείλει να είναι αναγνώσιμος και κατανοητός. Γιατί αλλιώς θα χάνουμε πάρα πολλά, θα έλεγα, δημοψηφίσματα εις βάρος μάλιστα της Ένωσης. Το πρόβλημα με την Ένωση είναι ότι δεν ομιλεί απευθεία με τους πολίτες. Οι υπουργοί συναντώνται, πολλές φορές όταν έρχονται εδώ στις Βεξέλλες συνεδριάζουν εκτός κοινοβουλευτικού εθνικού ελέγχου, δεν ελέγχονται από εμά, τα ψιλοβολεύουν χωρίς πρακτικά. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, κύριε Φερνάντες, για να κλείσουμε την υπόθεση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Ελπίζω να τις ε, στείλουν και γραπτός, ώστε να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε πολύ πριν τη διαμόρφωση της έκθεσης. Πάντως έχουμε χρόνο για να καταθέσουμε και τροπολογίες και να συντάξουμε και συμβαστικές τροπολογίες για το θέμα αυτό. Πάντως μετά από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση και μικρές αποκλήσεις. Ευχαριστώ. Si, alors nous allons suspendre pendant... Καλώς. Θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή τώρα και θα επανέλθουμε για την ανταλλαγή απόψεων με τον Μάριο Μότι, τον πρόεδρο της ομάδας ψηλό επίπεδο για τους ιδίους πόρους. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εγκαρδιότατα τον Μάριο Μόντι ως, με την ιδιότητα του ως πρόεδρου της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους. Θα μπορούσε κάλλιστα ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να έχει ίδιους πόρους. Περιμέναμε και λίγο νωρίτερα αυτή την ανακοίνωση της ομάδας υψηλού επίπεδου αλλά οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν. Πάντως χαίρομαι που ήρθε σήμερα στη συνεδρίασή μας ο Μάριο Μόντι για να μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά και το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις με τους ε, βουλευτές γιατί θα είναι ευκαιρία να συνεχίσουμε τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί για τους ίδιους πόρους ε, το αποφασιστικό βήμα θα εξαρτηθεί από τις αγαστές σχέσεις και την πλήρη σύμπνοια μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ ε, για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού ήταν ε, ουσιαστική σημασίας από την αρχή της εργασίας μας, της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ιδίους πόρους και βεβαίως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η υποστήριξη αυτή και για τη συνέχιση των εργασιών γιατί η πολιτική συνέχεια θα είναι δύσκολη. Θα είναι δύσκολη η συνέχιση μετά από τα δύο στάδια, το πρώτο στο οποίο, για το οποίο μας μίλησε ο Πρόεδρος και για το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δια, δια κοινοβουλευτική διάσκεψη τον Σεπτέμβριο και επίσης ε, η υποβολή της έκθεσης ε, πριν από το τέλος του 2016. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ανανέωση της υποστήριξης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την επανεπισήμανε την περασμένη εβδομάδα στο ψήφισμά του για ε, την ε, αναθεώρηση ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ε, ζητήσατε μία φιλόδοξη υποβολή έκθεση της ομάδας μου μέχρι το τέλος του έτους και παραμένουμε δεσμευμένοι στην υποβολή της έκθεσης αυτής εντός των προθεσμιών ε, με σεβασμό της εντολής την οποία λάβαμε από, τους, από τα τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι το γενναιόδωρο χρονικό διάστημα το οποίο δόθηκε στην ομάδα υψηλού επίπεδου για να εμβαθύνει το προβληματισμό της ήταν εποφελής για τρεις λόγους παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ ε, συνηθίσει εντός ε, ε, δύσκολων χρονοδιαγραμμάτων σε επίγουσες καταστάσεις να αποφασίζουμε ε, δεν ήταν η περίπτωση αυτή τη φορά. Μας δόθηκε λοιπόν ε, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος η δυνατότητα να έχουμε μία όριμη σκέψη. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα σε πολλά think tanks, ακαδημαϊκούς και πυρογνώμονες να συνεισφέρουν στον προβληματισμό αυτό. Και κατά τρίτον μας έδωσε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη ε, το εξελισσόμενο περιβάλλον και τις αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Να σας δώσω κάποιες ευκρινήσεις για τα δύο τελευταία σημεία που ανέφερα. Μεταξύ των πολλών ε, συνεισφορών που λάβαμε που είναι διαθέσιμες ε, στον ιστότοπο της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου υπάρχει η εξωτερική μελέτη εκ μέρους της ομάδας για το δυναμικό και τους περιορισμούς της αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η μελέτη αυτή μπαίνει σε λεπτομέρειες όχι μόνο για τα πιθανά ε, στοιχεία μεταρρύθμισης των ιδίων πόρων με νέα αξιολόγηση των ιδίων πόρων ε, και ε, μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των δαπανών. Επίσης παρουσιάζει ένα σύνολο πιθανών πακέτων ασυμφωνιών και πραγματεύεται τα ωφέλη τους. Επίσης, έχουμε ένα ευρύ πλούσιο φάσμα των ευρωπαϊκών οικονομικών από Γερμανούς εμπειρογνώμονες στις αρχές του χρόνου και καλύπτει μεγάλη κλίμακα ζητημάτων από τη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν απολογισμό του τι σημαίνει επικουρικότητα για τα οικονομικά, όπως για παράδειγμα για ε, έναν πιθανό φόρο ηλεκτρισμού ή φόρο αυτοκινούμενων οχημάτων. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να αναφερθώ στις διάφορες ε, συνεισφορές που λάβαμε. Ο προ, η, προ, η, προ, απερχόμενη Ολλανδική Προεδρία μας υποστήριξε πάρα πολύ και συνεισέφερε πολύ, ειδικότερα ως προς τη σχέση μεταξύ της αναθεώρησης ε, της σχέσης μεταξύ εσόδων και εξόδων, που ξέρουμε ότι είναι οι δύο όψεις της ίδιας πρόκλησης, προκειμένου ο ε, προϋπολογισμός της Ένωσης να είναι πιο επαρκή στο μέλλον. Όλες αυτές ε, οι συνεισφορές ήταν πάρα πολύ τιμές ε, λόγω του ε, δύσκολου ε, κλίματος με έντονες αναταράξεις που συνεχίζεται ακόμη. Όταν αρχίσαμε τη δουλειά μας κατά το πρώτο ήμιση του 2014, η η διάθεση ε, δεν ε, ήταν να συζητήσουμε ουσιαστικά ζητήματα όπως η λειτουργία του ενωσιακού προϋπολογισμού ή ε, οι ευθύνες τις οποίες θα έπρεπε να περιέχει αυτός. Η συνεχιζόμενη όμως οικονομική κρίση και η μενόμενη προσφυγική κρίση άλλαξαν την ε, πορεία μας γιατί είχα, είχε αποτέλεσμα ε, σε μεγάλο βαθμό ε, στις διάφορες πολιτικές μας αν η ημερομηνία για την υποβολή της έκθεσής μας είχε οριστεί για παράδειγμα κατά για τα μέσα του 2015 θα ήταν τελείως διαφορετική η έκθεση, πολύ πιο ε, ρουτίνας, ε, ε, με περισσότερα περιθώρια ε, βελτίωσης, όμως είχαμε την Ε, το όφελος, ε, για να το πω έτσι, πολλών ε, παράλληλων κρίσεων που μας επέτρεψαν, γι' αυτό ήταν εποφελής, να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο ως προς την θεμελιώδη και εκβάθρων μεταρρύθμιση του ενωσιακού προπολογισμού, ο πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό πλέον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό ε, και δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό αν δεν είχαν εμφανιστεί ε, τόσο απρόπτα όλες αυτές οι κρίσεις και οι προκλήσεις. Κατά το Κατά τον τελευταίο χρόνο οι εθνικές κυβερνήσεις, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ ξανά δεν είχαν υποχρεωθεί να ε, γυρίσουν πίσω στην ε, ιδέα ε, του δημοσίου αγαθού της Ένωσης που είναι κάτι το οποίο είχε παραγνωριστεί ή είχε τεθεί στο παρασκήνιο των πολιτικών των συζητήσεων για τις πολιτικές κατά τα τελευταία χρόνια ε, ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε στο πλαίσιο της προστιθέμενης αξίας, όμως ε, οι τρόποι εφαρμογής αυτής της προστιθέμενης αξίας είχαν κάπως ε, χαθεί, όπως και η ιδέα του δημόσιου αγαθού στις κοινωνίες μας, οι οποίες είχαν ως γνώμονα κυρίως τη μεγιστοποίηση του ε, συμφέροντος του ιδιώτη, του καταναλωτή και τη μείωση της φορολογικής πίεσης όταν αυτό ήταν δυνατόν, ε, ενώ τα δημόσια αγαθά και ειδικότερα τα δημόσια αγαθά που ευτυχώς ή δυστυχώς μπορούν να παραχθούν αποτελεσματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, επανέλθει στο προσκήνιο. η δυστυχως μπορουν να απαραχθούν αποτελεσματικα σε επιπεδο ευρωπαικης ενωσης εχουν επανελθει στο προσκηνιο η η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια που είναι όλο και περισσότερο δύσκολο να τις αντιμετωπίζει κανείς ξεχωριστά, η ποιότητα του περιβάλλοντος ε, με παγκόσμια συμφωνία που επετεύχθη στην COP21 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε ε, ηγετικό και πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Όλες αυτές οι προκλήσεις για, από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών, των πολιτών μας και όλο και περισσότερο θα εξαρτάται ε, στο μέλλον ε, σε σχέση με αυτό που πιστεύαμε πριν από 12 μήνες. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να ε, κάνει κανείς καμία πολύ λεπτομερή εξέταση για να καταλάβει ότι σήμερα δεν επαρκεί ο προπολογισμό της Ένωσης για να εκπληρώσει τα καθήκοντα αυτά και ελπίζουμε ότι θα πιέσουμε για φιλόδοξη μεταρρύθμιση ε, του ενωσιακού προπολογισμού. Είναι και διαφορετικό αυτό το οποίο ε, ε, θεωρεί το φιλόδοξο πέρσι είναι πλέον ε, ουσιώδες για την ε, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα έσοδα και τις δαπάνες. Γι' αυτό έχουμε κατά κάποιο τρόπο αυξήσει το ελάχιστο όριο των ε, φιλοδοξιών μας. Ε, εμείς επικεντρωνόμαστε στον τομέα των ε, εσόδων, γι' αυτό θα υποβάλουμε κυρίως την έκθεση, όμως επισημαίνουμε ότι και οι δύο μεταρρυθμίσεις πρέπει να λάβουν χώρα παράλληλα. Υπάρχουν κάποιες ενδεχόμενες νέες πηγές εσόδων που θα μπορούσαν να προέρχονται από τις πολιτικές και να παρέχουν χρήματα στον ενωσιακό προϋπολογισμό και να δημιουργήσουν κίνητρα για νέε ευρωπαϊκές πολιτικές, ειδικότερα ε, στον, ε, στο περιβάλλον, τι μεταφορέ, την οικονομική σταθερότητα μεταξύ άλλων και επίσης έσοδα μπορούν να προκύψουν από κάποιε πολιτικέ της Ένωσης που μπορεί να είναι σημαντικές αλλά δεν τροφοδοτούν τον προπολογισμό της Ένωσης και ανακατανέμονται σε ε, στους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, μέσω περίπλοκων υπολογισμών. Όλα αυτά πρέπει να τα ε, εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Σε αυτή τη φάση έχουμε διεξοδικά συζητήσει όλα αυτά τα ζητήματα και το επόμενο ορόσημο ε, της δουλειάς μας θα είναι να συζητήσουμε κάποια από αυτά πιο σημαντικά με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, με ε, εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, λίγο παραπάνω σε αυτήν ε, την διάσκεψη, η οποία ε, είναι πολύ σημαντική από πολιτικής και ψυχολογικής απόψεως, γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε τα εθνικά κοινοβούλια, αυτός είναι ο στόχος, στις στις εργασίες μας ε, που έχουν δρομολογηθεί. Είπατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, ότι στο παρελθόν έχουν παραγνωριστεί τα Εθνικά Κοινοβούλια στην αρχική αυτή φάση των συζητήσεων και συμμετείχαν μόνο όταν υπήρχε κάποιος επίσημος ρόλος για αυτά, όπως για παράδειγμα όταν έπρεπε να ληφθεί απόφαση ή να επικυρωθεί απόφαση για τους ιδίους πόρους. Το ε, γεγονός ε, ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου είναι διοργανική, και παρά το γεγονό ότι δεν είναι πλέον προνόμιο των εθνικών κοινοβουλίων, ε, είναι ε, να ε, διευρύνουμε τη συζήτηση. Και σας είπα προηγουμένως ότι αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Ελπίσουμε ότι αυτή η διάσκεψη θα δώσει την, ε, το απαραίτητο βήμα στα εθνικά κοινοβούλια για να αποκτήσουν μια κυριότητα αυτή της, της συζήτησης για την μελλοντική οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες των κοινοβουλίων στην τελική μας έκθεση. Και γι' αυτό ε, το λόγο τρία πάνελ έχουμε προβλέψει. Έχουμε στείλει ένα σημείωμα στους ε, συμμετέχοντες για να τους εξηγήσουμε ε, τα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Τρεις θεματικές ενότητες όπως και τα πάνελ. Το πρώτο ποιο ρόλο ε, πρέπει να διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της Ένωσης ε, στα δημόσια οικονομικά της Ένωσης. Ε, επίσης, δεύτερον, νέοι πόροι εσόδων, ε, τι λειτουργεί και τι θα έπρεπε να αλλάξει. Και τρίτο πάνελ, ε, καλύτερη συνοχή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ του προπολογισμού της Ένωσης και των εθνικών προπολογισμών, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα, που θα είναι βέβαια μία σαφής πρόσκληση προς τους συναδέλφους σας από τα Εθνικά ε, Κοινοβούλια. Ξεχνάω ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα έχουμε λοιπόν έναν πάρα πολύ ε, συγκεκριμένο διάλογο. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι βεβαίως ε, ε, ουσιώδης. Εσείς, κύριοι και κυρίες ε, ε, ευρωβουλευτές ε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο όπως και οι υπόλοιποι ομιλητές το πάνελ συμπεριλαμβάνει και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και μέλη της ομάδας υψηλού επίπεδου που θα κάνουν μια εισαγωγή σε κάθε θεματική ενότητα. Αν θέλετε να συμμετέχετε, έχουμε έναν ε, ιστότοπο για αυτό το σκοπό, όπου τα έγγραφα που ε, συζητήθηκαν από την ομάδα υψηλού επίπεδου σε όλες τις συνεδριάσεις, όπως επίσης και ακαδημαϊκά, ε, ακαδημαϊκά, έγγραφα, έγγραφα από τους ακαδημαϊκούς και ε, ανακοινοθέντα τύπου μπορείτε να τα βρείτε, υπάρχουν σε αυτόν τον ειδικό ιστότοπο. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα κύριε Πρόεδρε για το πώς μπορεί να συνεχίσει η ομάδα υψηλού επίπεδου από τη στιγμή που θα έχει υποβάλει την τελική της έκθεση. Θα ήθελα να αναφέρω ότι θα έχουμε ακόμη μερικές συνεδριάσεις το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να συζητήσουμε το περιεχόμενο ε, των εκθέσεων, της έκθεσης ε, σε με περισσότερη λεπτομέρεια και αυτό βεβαίως θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από ε, την ανταλλαγή απόψεων που θα λάβει η χώρα στην διάσκεψη. Ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου να υποβάλουμε την έκθεσή μας ή μέσα Δεκεμβρίου Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα ε, συστάθηκε ε, από ε, τα τρία όργανα από τους τρεις προέδρους ε, στο Στρασβούργο και συνεπώς σε αυτούς θα απευθύνεται η έκθεση ε, και νομίζω ότι θα ήταν ευγενικό ε, και προς το πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι μόνο τον προεδρεύοντα να το υποβάλουμε και βεβαίως θα υποβάλουμε απευθείας και σε εσά τη χρονική στιγμή που θεωρείται κατάλληλη. Και επίσης Ήρθαμε σε επαφή και με τις υπηρεσίες σας, ε, ώστε κατά τις επόμενες ημέρες ε, να υπάρξει μία ε, απόφαση πότε ακριβώς θα κάνουμε την υποβολή της έκθεσής μας σε εσά, σε ποια ημερομηνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται από την εντολή της ομάδας υψηλού επίπεδου, πρέπει να αξιολογήσει τα ε, πορίσματα και να αποφασίσει κατά πόσο θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τους ιδίους πόρους. Αφού λοιπόν ε, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τα ε, τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μας εμπιστεύθηκαν αυτό το δύσκολο έργο ε, η εξουσία θα μεταφερθεί, ε, είναι ακόμη, είχε ακόμη το μονοπόλιο της νομοθετικής πρότασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποφασίσει εκείνη αν πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τους ιδίους πόρους. Η συνέχιση ε, στους, ε, στα άλλα όργανα θα είναι απόφαση των οργάνων αυτών και Είμαι πεπισμένος ότι θα ε, συνεισφέρεται ε, και μετά ε, την υποβολή της έκθεσης για την... Για τον... Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε τη συζήτηση θέτοντας δύο προβλήματα τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια πάλι προβλήματα τα οποία νομίζω είναι και δικά σας, είναι τμήμα των ανησυχιών στην, στο ψήφισμά σας την προηγούμενη εβδομάδα. Τα δύο αυτά θέματα έχουν συζητηθεί από την ομάδα μου εξαντλητικά θα έλεγα και θα αποτελέσουν τμήμα και της τελικής μας παρουσίασης. Το πρώτο από τα θέματα αυτά έχει σχέση με τον σύνδεσμο ανάμεσα στις πηγές εσόδων και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο θέμα είναι μια βασική ανησυχία την οποία έχετε και εσείς και εμείς και αφορά την αύξηση του αριθμού των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση. Για το πρώτο πρόβλημα, για τη σχέση ανάμεσα στις πηγές εσόδων και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται θα έλεγα της ευρύτερη συζήτηση για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι μια έννοια η οποία δεν είναι εύκολα αριθμητικά προσμετρήσιμη. Πάντως τα ωφέλη για την ε, ε, ενιαία αγορά είναι δεδομένα. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, πολύ συχνά ε, εκτιμούμε ε, κάποια προβλήματα ή κάποια στοιχεία μάλλον τα οποία ε, είχαμε, αλλά ξαφνικά τα χάνουμε ή κινδυνεύουμε να τα χάσουμε και τότε καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία τους. Νομίζω ότι η σημασία την οποία έχει η ενιαία αγορά έχει πλέον υπογραμμιστεί ιδιαίτερα μετά από αυτό το οποίο έγινε μετά από την αποχώρηση ενός κράτους μέλους. και το οποίο λέγει ότι θέλει να συνεχίσει να ωφελείται από την ενιαία αγορά. Αυτό δείχνει ακριβώς τι σημαντικές δυσκολίες θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις ε, προϋποθέσεις και στις συνθήκες έτσι ώστε μια χώρα που δεν είναι πλέον μέλος να μπορεί να συνεχίσει να ωφελείται από την ενιαία αγορά. Ανεξαρτήτως του αν αυτό το κράτος μέλος ή τέος κράτος μέλος έχει προκαλέσει εν πολλής ε, την δημιουργία αυτού του κοινού αγαθού, το οποίο επαναλαμβάνω ονομάζουμε ενιαία αγορά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι δυσκολίες δεν θα εμφανιστούν στο σύνολο των διαπραγματεύσεων, πάντως ε, απαιτείται δυστυχώς μερικές φορές να υπάρξει ένα τράνταγμα μεγάλο για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα θετικά τα οποία έχουμε. Τα ωφέλη λοιπόν από την ενιαία αγορά είναι κάτι το σημαντικό. Σε επίπεδο δημοσιονομικό βέβαια δεν είναι θέμα κοινοτικών πολιτικών, είναι θέμα κοινών κανόνων και όχι προγραμμάτων στα πλαίσια των οποίων δαπανώνται ε, κάποιες πιστώσεις. Και είναι κάτι το οποίο δεν συνδέεται και άμεσα με τις ε, εθνικές εισφορές ε, αν δούμε μια χώρα ας πούμε η οποία δεν είναι κράτος μέλος, η Νορβηγία και η οποία έχει έρθει πολύ στην επικαιρότητα περιέργως τελευταία, ε, συμμετέχει στην ενιαία αγορά και συμμετέχει σε ορισμένες επιλεκτικά πολιτικές, συνεισφέρει στον προπολογισμό η χώρα αυτή πάνω από δύο φορές από τις προβλεπόμενες ε, καταρχάς δαπάνες. Αυτό δείχνει ότι η συμμετοχή στην ενιαία αγορά είναι πολύ περισσότερες ε, ε, από ό,τι φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο, σε επίπεδο μιας πρώτης ανάγνωσης. Και δεν έχουμε να κάνουμε με μια ρομαντική χώρα η οποία ξοδεύει χωρίς να σκέφτεται. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μου θεωρεί ότι ακριβώς πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα λεγόμενα κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, τα οποία ποσοτικά δεν είναι άμεσα προσμετρήσιμα, αλλά είναι επαρκές θεμέλιο ε, για να ε, μειωθεί η σύγκρουση που πολλές φορές έρχεται στην επικαιρότητα σχετικά με τις εθνικές εισφορές. Υπάρχουν ε, λοιπόν κοινέ ευθύνε γύρω από τα θέματα αυτά. Ε, υπάρχει το θέμα σαν παράδειγμα της ασφάλειας ε, και της κάλυψης των αναγκών για την ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν αποτελεί συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διάφορες χώρες ε, εφαρμόζουν μέτρα γύρω, στον, από τον τομέα της ασφάλειας ε, και ζητούν ταυτόχρονα εξαιρέσεις των ποσών αυτών από τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του χρέους και του ελλείμματος κτλ. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα όπως θα τα ήθελαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μια σημαντική αμυντική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οποία οι πολίτες υποστηρίζουν με συστηματικό θα έλεγα τρόπο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό, αν και δεν θα συμφωνούσαν όλες οι χώρες μέλη. Και η συμπληρωματικότητα εδώ με, τη, με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής παρέμβασης θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο κατάλληλη θα έλεγα κατανομή των δράσεων. Ίσως να υπάρχουν λοιπόν κάποιες λύσεις έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον τομέα των εσόδων δημιουργούντας ιδίους πόρους οι οποίοι να συνδέονται με έναν στόχο, μια προτεραιότητα, μια πολιτική. Αυτό το έχουμε κάνει στο παρελθόν, το έχουμε εξετάσει εννοώ, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσιονομική σταθερότητα, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ό,τι άπτεται τη φορολογίας γενικά, το λεγόμενο FAT, περιβάλλον, καταπολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών, φόρος ε, του άνδρακα, ε, κατανομή των εσόδων, ένας επιπλέον πιθανός ίδιος πόρος, αύξηση των επενδύσεων στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ακριβώς ad hoc πόρων, ο κατάλογος τον οποίο σας έδωσα δεν είναι φυσικά εξαντλητικός και δεν είναι ο βασικός μας στόχος, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε είναι ότι το θέμα των εσόδων είναι κάτι που μπορεί να πετύχει στους στόχους, να βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους, όπως και η δημοσιονομική ας πούμε πολιτική και έτσι να καταστεί και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πιο σαφής. Και τώρα έρχομαι στο δεύτερο σημείο το οποίο είπα ότι πρέπει να θέσω. Οι βασικές ανησυχίες γύρω από, την, από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μέσων που χρηματοδοτούνται ad hoc. Ε, δεν χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πόση καινοτομία και πόση ευελιξία μπορούμε να ανεχθούμε έτσι ώστε να μην τεθεί σε απειλή η αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού και η δημοκρατική του νομιμοποίηση. Ε, κάποια κατεπήγοντα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί με λύσεις ad hoc, ε, μέσω δημιουργίας trust funds, ε, μέσω του μέσου για τους πρόσφυγες στην Τουρκία κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κράτη-μέλη έδειξαν ότι έχουν την βούληση να δώσουν δύο δις επιπλέον το 16 και 17 και τα ποσά αυτά να περάσουν από τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς και ταυτόχρονα έτσι να ε, ε, υπάρξει και η ομοφωνία που απαιτείται. Αυτό δείχνει ότι ένα ευέλικτο και συντονισμένο ευρωπαϊκό επίπεδο προόδου μπορεί να ευρεθεί κάτι, όταν είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν συνειδητοποιεί πλήρως και τα αρνητικά σημεία αυτών των εφάνταστων δημιουργικών λύσεων. Ε, μπορεί να σας δώσω εδώ, θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Ε, τα μέσα αυτά δίδουν κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν είναι ικανοποιητικά σε επίπεδο δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν πράγματι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι επαρκή ε, όταν βλέπουμε ότι κάποια κατεπήγοντα θέματα σιγά σιγά διαμορφώνονται σε διαρθρωτικά προβλήματα γιατί είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων. Αυτό που ονομάζουμε μερικές φορές ε, κατεπήγον είναι κάτι το οποίο μας αποκαλύπτει τελικά ένα μονιμότερο πρόβλημα. Και γίνεται ουσιαστικά ένα διαφορετικό φαινόμενο. Όπως είπα, τα κατεπήγοντα αυτά απαιτούν μερικές φορές στρατηγικούς τρόπους αντιμετώπισης. Είναι σαφές επίσης ότι αυτές οι ad hoc, οι επιτούτου λύσεις, επιλέγονται για συγκεκριμένους λόγους κάθε φορά. Όταν απαιτείται ένα ψηλότερο επίπεδο ιδίων πόρων και πληρέστερο επίπεδο ιδίων πόρων που θα καθιστούσε τις επιμέρους αυτές λύσεις ε, ε, περιτές. Από πλευράς κοινοτικού προϋπολογισμού θα πρέπει κάποιες, ε, θα έλεγα, σύγχρονες εφάνταστες λύσεις να συμβαδίζουν με την απαραίτητη πάντα μορφή δημοκρατικού ελέγχου υπάρχει ένα τμήμα των εσόδων προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θεωρείται ίδιος πόρος και έχει τον όχι και πολύ ελκυστικό τίτλο Other Revenue, άλλα έσοδα. Εδώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες από την πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια στην παρούσα φάση δεν παρέχουν τις δυνατότητες που θα επιθυμούσαμε. Αυτό το οποίο έχει σημασία βέβαια είναι ότι τέτοιου είδους έσοδα δεν ακολουθούν την διαδικασία των ιδίων πόρων, αλλά δευτερογενές δίκαιο. Ένα παράδειγμα είναι σαν παράδειγμα είναι ε, τα πρόστιμα για την παραβίαση του ανταγωνισμού στα πλαίσια διαπίστωσης καρτέλ όπως επίσης ε, τα επιπλέον ποσά τα οποία μπορεί να προέρχονται από παραβιάσεις των κανόνων εκπομπών νέων οχημάτων όπως επίσης και μέτρα φορολογικού τύπου στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας άρθρα 192 και 194 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιου είδους μέτρα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως ακόμα θα πρέπει να τεκμεριωθούν πρώτα σε σχέση με την χρησιμότητά τους και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τα τέλη αυτά, τα πρόστιμα αυτά, οι διαδικασίες αυτές πολλές φορές χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα μπορούσαν να είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των κοινοτικών πολιτικών στο μέλλον. Σας ζητώ συγγνώμη διότι πραγματικά μακρηγόρησα. Ήξερα κύριε Πρόεδρε, είχα πληροφορίες ότι η Επιτροπή σας θεωρούσε ότι είναι αναγκαίο, ότι είναι χρήσιμο να προσπαθήσει να ανακτήσει λίγο ε, την γνώση που απαιτείται ε, για να κατανοηθούν οι προσπάθειες που κάνουμε εμείς σαν ομάδα. Και νομίζω ότι τώρα σας έδωσα ίσως και κάποια επιπλέον στοιχεία να είστε ενήμεροι και να κάνετε την κριτική που απαιτείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπετε και από τα χειροκροτήματα πώς, ε, με ποιο τρόπο γίνεται δεκτή η παρουσίαση. Περιτεύουν τα λόγια. Όλα αυτά που μας ε, εκθέσατε ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες μας και στις αδημονίες μας. Δημοσιονομική ενότητα. Εγώ θα έλεγα και ε, εύληπτο προϋπολογισμό ευανάγνωστο προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό που θα εξυπηρετεί μια κοινότητα ε, αλλά όταν είναι δυσανάγνωστο ο όταν τα μέλη δεν μπορούν να το καταλάβουν, είναι ευάλωτος. Γι' αυτό θα πρέπει να καταστήσουμε εύληπτο τον προϋπολογισμό για τους Ευρωπαίους πολίτες, κατανοητό. Θα πρέπει οι συμπολίτε μας να αντιληφθούν αυτή την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η προστιθέμενη αξία είναι τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Τότε θα αγγίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την καρδιά των Ευρωπαίων. Αλλά χρειάζεται γι' αυτό δημοσιονομική ενότητα. Είναι ένα ολόκληρο στερέωμα, ένα συνδυασμό και θα πρέπει σε αυτό το στερέωμα να προκαλέσουμε τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang ένα στερέωμα, ίσως ένας αστερισμός, αλλά μέσα σε νύχτα, σε μαύρη, ζωφερή νύχτα. Ναι, αλλά δεν θα αργήσει και το φως που θα φωτίσει αυτή τη νύχτα. θα δώσω το λόγο τώρα στους συζητητές. Ο Αλένα Λαμασούρα όμως που συμμετέχει αυτό στην ομάδα υψηλού θα μπορούσε πρώτα να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Ε, είχα το προνόμιο να είμαι ταυτόχρονα αναπληρωτής, αναπληρωματικό μέλος της ε, Επιτροπής Προπολογισμών και μέλος της ομάδας υψηλού επίπεδου, στην οποία προεδρεύει ο κύριος Μότη. Θα ήθελα να τη φόρο τιμή ε, στον κύριο Μόντι και να σας διαβεβαιώσω ότι η ομάδα του τηρεί την εντολή που της ανατέθηκε και με μία συνενετική μέθοδο καταφέρει να παρουσιάσει τα πράγματα. Βέβαια για το σκοπό δεν υπάρχει απόλυτη συνένεση. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μόντι και όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής ψηλεπέτα το γνωρίζουν, ε, οι εξέλιξη της τελευταίας διετίας επιβεβαιώνουν αυτά που είχε πει η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι είχε δικαιολογήσει την πρότασή της για τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση του συστήματος ιδιών πόρων. Είχε πει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο προπολογισμό και το πλαίσιο, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 είναι απολύτω ακατάλληλα για να ανταποκριθούν στι νέε ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη και το λέω ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ανακύπτει το ερώτημα. Ε, εξακολουθεί να ισχύει ε, αυτό, αυτή η καταλληλότητα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί συνεχίζονται τα πρόβλεπτα και πολύ πιθανό μετά την επταετία αυτή το τοπίο να έχει αλλάξει ριζικά. Εξακολουθεί λοιπόν να είναι κατάλληλος αυτός ο προγραμματισμός. Και μήπως ε, θα πρέπει να επανανομιοποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε εκ βάθρων τον κλασικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γιατί Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που όπως είπατε έχουμε έναν αστερισμό ή ένα στερέωμα προϋπολογισμών διακρατικών που ε, θεσπίζονται για να χρηματοδοτήσουν τις νέες ανάγκες και στον κοινοτικό προϋπολογισμό, στον ενωσιακό προϋπολογισμό, όταν χρειαζόμαστε πόρους για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχέδιου Juncker, την ε, μετατροπή ε, της Frontex σε ένα πραγματικό οργανισμό ελέγχου του εξωτερικού συνόρων ή για να χρηματοδοτήσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία με την Αφρική ή να περιορίσουμε τις εκπομπές του άνθρακα. Ουσιαστικά για τη χρηματοδότηση προσφεύγουμε σε αυτό που αποκαλέσατε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και τα μόνα στοιχεία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προστατεύουμε τελευταία ε, αιτία είναι η τα προκαθορισμένα κονδύλια, το 80% δηλαδή του προπολογισμού που προορίζονται για τα κράτη-μέλη. Οπότε δεν υπάρχει πια, δεν έχει απομείνει ενωσιακό προπολογισμό. Ας μην βαφκαλιζόμαστε. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να το δηλώσουμε. Δεν υπάρχει πια ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και το Brexit θα μα υποχρεώσει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, αρχής γενομένης από το GNA. Γιατί από τη στιγμή που δεν θα έχουμε το, Ευρωπαϊκό, το, την, το Βασίλειο στην Ένωση, δεν θα έχουμε και την επιστροφή. Και ούτε για, το, για τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε για τι υπόλοιπε επιστροφέ. Γιατί οι υπόλοιπε επιστροφέ αντλούσαν την ομοποίησή του από την επιστροφή προ τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε εκεί θα έχουμε πολύ σημαντικό επιχείρημα. Άλλη έμεση συνέπεια του Brexit είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα τους επόμενους μήνες και χρόνια θα αναλυφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες για νέες πολιτικές στα πλαίσια του τωρινού προϋπολογισμού, ίσως μέσω της νομικής ε, μορφής της ενισχυμένης συνεργασίας. Και μάλιστα η χθεσινή κοινή δημόσια κρόαση μεγάλης εμβέλειας έδειξε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι και πολύ υπέρ μια δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνη, ενό προπολογισμού τη Ευρωζώνη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αναλυφθούν άλλε πρωτοβουλίε, πολύ πιθανόν αμυντικού χαρακτήρα, για να εξετάσουμε και εκεί τι πολιτικέ μα. Και στα θέματα τη ενέργεια, ίσω θα χρειαστεί να ε, διαρωτηθούμε για τη χρήση των πόρων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Οπότε θα πρέπει να δικαιολογήσουμε τις μας και ίσως χρειαστεί να επανεφεύρουμε τον ενωσιακό προϋπολογισμό και ίσως χρειαστεί να τεθεί ένα αμφιβόλο ή να χρειαστεί και επαναπροσδιορισμός του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σε αρχές ε, Σεπτεμβρίου θα συναντηθούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και στο ισχύον πλαίσιο ευρωσκεπτικισμού, έξαρσης του ευρωσκεπτικισμού και αυξανόμενων αφιβαλιών ε, ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομίζω ότι το μόνο μέσο που έχουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι να αποδείξουμε εμπράκτος με παραδείγματα και με αριθμητικά στοιχεία ότι αν εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας και αν εμείνουμε στις κοινοτικές αρμοδιότητες της Ένωσης, ένα ευρώ που ξοδεύουμε σε κοινοτικό επίπεδο θα μας επιτρέψει να εξοικονομήσουμε ε, ένα σημαντικό τμήμα του τη φορολογική επιβάρηση προς τους φορολογωμένου και να εξοικονομήσουμε και κονδύλια σε εθνικό επίπεδο. Και ελπίζουμε ότι με τον παρέμβαση ευρωπαϊκή Ένωση θα ελαφρύνουμε την συνολική φορολογική επιβάρηση των συμπολιτών μας και όχι να την ενισχύσουμε. Πάντως ε, είμαι οργισμένος, εξοργισμένος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημείο αυτό. Γιατί πάνε 18 μήνες που στα πλαίσια κυρίως της ομάδας υψηλού επίπεδου, αλλά και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ζητούμε εντόνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό το εγχείρημα. Ή τουλάχιστον να το αναθέσει στο ελεγκτικό συνέδριο ή στα δίκτυα εθνικών ελεκτικών συνεδρίων. Αλλά ούτε ακόμα έχει, δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή η στα δικτυα εθνικων ελεγκτικων συνεδριων αλλα ουτε ακομα δεν εχει ξεκινησει καν αυτη η διαδικασια Και αν δεν το παρουσιάσουμε αυτό θα μας συντρίψουν με τα επιχειρήματά τους στα Εθνικά Κοινοβούλια κατά την παρουσίαση των προτάσεων. Και εν ώψη της συνάντησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια, καλό θα ήταν οι Ευρωβουλευτές να προσπίσουν ένα ευρωπαϊκό όραμα. Δεν έχουμε όλοι κοινή αντίληψη για το ευρωπαϊκό όραμα, για τη μορφή που θα πρέπει να έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά νομίζω ότι όλοι, και αυτή είναι η πολιτική μας προστιθέμενη αξία, έχουμε μία, ένα όραμα για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και μια και όλο και περισσότερο θα προβάλλονται εθνικές ή εθνικιστικές απόψεις ε, στις συζητήσεις, θα πρέπει εμείς να προσπίσουμε το ευρωπαϊκό όραμα, την ευρωπαϊκή προοπτική. Να και είμαστε οι αμύντορες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Προοπτικής. Ο κύριος Λεβαντός και απουσιάζει, ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ιδιαίτερο ευτυχής ε, που άκουσα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μόντι στο εσωτερικό ενός πλαισίου θα έλεγα που, όπου ακούγονται μόνο κλαφμοί, οδυρμοί και ευρωσκεπτικισμός Αυτά τα οποία μας είπε ήταν παρηγορητικά. Βλέπω ότι πιστεύετε ότι η κρίση είναι ευκαιρία όχι για να παρετηθούμε, αλλά για να ανυψώσουμε το επίπεδο των απαιτήσεών μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή στάση. Με χαρά σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι αυτή στιγμή βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι προκλήσεις. Θα προσανατολιστείτε σε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού και σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτό που είπατε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να σταθεί κυρίως σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά αγαθά, κοινά αγαθά, Κοπέρνικος και η επανάστασή του. Ένα από τα βασικά αγαθά αυτά δεν είναι το πιο ακριβό άλλωστε. Αναφερθήκατε στην ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι αυτή που επιτρέπει αν θέλετε τα περισσότερα κέρδη και επιτρέπει επίσης την Ορβηγία να πληρώνει για την συμμετοχή διότι το θεωρεί χρήσιμο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρώτο μάθημα στο οποίο μπορεί να καταλήξει κανείς. Ένα δεύτερο παράδειγμα Είπατε ότι το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εξωτερική αλλά και την εσωτερική. Η εσωτερική ασφάλεια δεν είναι ε, θέμα δισεκατομμυρίων μόνο, αλλά είναι και θέμα ευφυΐας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών, εάν ανταλλάσσουν σωστά τις πληροφορίες τους, εάν υπάρχουν διαδικασίες ε, οι οποίες αντίθετα από τις σημερινές όταν εντοπίζουν κάποιον μπορούν να το ανακοινώνουν αυτό στις υπηρεσίες των άλλων χωρών. Δεν θα γίνουν αυτά τα οποία δυστυχά, δυστυχώς έγιναν με τον κύριο Αμπτελσλάμ και άλλους το τελευταίο καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι η λογική σας είναι ιδιαίτερα θετική. Μία ερώτηση μόνον. Ίσως να διερμηνεύω λανθασμένα αυτό το οποίο θελήσατε να πείτε. Στην ουσία προσπαθείτε να βρείτε κάποιους πόρους οι οποίοι να χρησιμοποιούνται άμεσα στα πλαίσια κάποιων πολιτικών. Αντίθετα δηλαδή από αυτό που γίνεται σε πολλούς προϋπολογισμούς όπου ε, τα χρήματα τα οποία θα έλεγα έχουν σαφή προσανατολισμό εξ αρχής μπορούμε εν πάση περιπτώσει να εντοπίσουμε συγκεκριμένους σπόρους ε, για συγκεκριμένες δράσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει ενδιαφέρον σε δημοσιονομικό επίπεδο. Και μία επιπλέον ερώτηση. Υπογραμμίσατε ιδιαιτέρως στην παρουσίασή σας την ε, διάσκεψη της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Και αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε, αυτό το οποίο αναζητείτε ε, είναι να δείτε αν υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ε, και για τον τομέα των ιδίων πόρων. Δεν θέλετε να συζητήσετε με τα κοινοβούλια την καταλληλότητα ή μη συγκεκριμένων ιδίων πόρων. Η αίσθησή μου είναι ότι ανοιχνεύεται το έδαφος για να δείτε αν θα υπάρξει μια άρνηση ή μια αποδοχή ε, του προσανατολισμού τον οποίο εσείς αναφέρατε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω προς το παρόν κύριε Μόντι, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Έχουν ζητήσει άλλοι τρεις συνάδελφοι το λόγο, θα ήθελα παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί σε πολύ λίγα λεπτά, σε έξι λεπτά, διευρύνουμε τη συνεδρίασή μας με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να δούμε τι συμβιβαστικές λύσεις μπορούμε να βρούμε ε, με τις τροπολογίες Μπερές και Μπόγκε. Ο κύριος Ντονανό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την ελπίδα την οποία μας δίδετε με αυτά που είπατε. Ευχαριστώ για την έννοια επίσης του κοινού αγαθού. Ε, χρειάζεται χρόνος βέβαια για να το πετύχουμε αυτό ε, και πράγματι είναι κατεπήγον το θέμα Και μιας και η έκθεση αυτή οδηγεί την Επιτροπή να κάνει νέες προτάσεις, πιστεύετε ότι οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν ομόφωνα δεκτές ή θα πρέπει να ε, στραφούμε σε, μια, σε έναν πυρήνα κρατών ή και στη ζώνη ευρώ. Η κυρία Γουάρια Ζαμπάλα, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι ήταν ε, ελπιδοφόρο και ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εργασίες της ομάδας υψηλού επίπεδου. Μας είπατε ότι καταρχάς εμείς μιλάμε για συγκεκριμένες φιλοδοξίες τις οποίες μπορούμε να έχουμε και πέρα από τις φιλοδοξίες αυτές πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το θέμα είναι επίγον. Βέβαια με ανησυχεί το ότι τα κράτη-μέλη δεν παρακολουθούν την κατάσταση αυτή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εμείς το κάνουμε. Εμείς συζητήσαμε πριν λίγο καιρό για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υπουργούς και δεν είδαμε να υπάρχει μια θέληση, να υπάρξει μια λύση αλλά και μετά από αυτά που είπε ο κύριος Λαμασούρ στον τομέα των προσφύγων, της ενέργειας, της καταπολέμησης, της τρομοκρατίας. Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σωστά. Δεν είναι όλα χρήματα βέβαια, αλλά τα χρήματα είναι απαραίτητα και απαιτείται αύξηση των ιδίων πόρων. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Συμβούλιο. Ε, έστω και μέσω αυτού του ελάχιστου κοινού παρανομαστού. Θα πρέπει έστω να καταλήξουμε στην λιγότερο φιλόδοξη των απαντήσεων και ελπίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες προέρχονται από την ομάδα υψηλού επίπεδου να μην είναι ο κοινό ελάχιστος παρανομαστής αλλά ο μέγιστος δυνατός. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μπορέσουμε το σύνολο αυτό των εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πόρων ε, να το εξετάσουμε όπως επίσης και για την Ευρωζώνη άλλωστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν 1,5 χρόνο ήσασταν εδώ λέει ο κύριος Βιώτη και είχατε πει ότι η παρουσίασή σας τότε στην ουσία ήταν μια φεά παρουσίαση θεά διότι δεν υπήρχαν πάρα πολλά σημεία ελπίδας. Ενώ τώρα μας δώσατε μια έκθεση κάπως πιο έγχρωμη θα έλεγα και ελπίζω ότι και η τελική σας έκθεση θα είναι και αυτή επαρκώς έγχρωμη. Να μου επιτρέψετε εδώ να σας συγχαρώ επίσης γιατί βάλατε online και τα έγγραφα εργασίας τα οποία χρησιμοποιείτε. Είναι ε, φυσικά πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι φυσικά όλοι οι πολίτες εμπειρογνώμονες στα θέματα των ιδίων πόρων. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή. Τώρα δεν θα ήθελα να, παρι, να μακρηγορήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα έφεσαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Πάντως η προσπάθεια την οποία θα πρέπει να κάνουμε από το μήνα Δεκέμβριο και μετά είναι να ξεφύγουμε λίγο από το τεχνικο-οικονομικό χαρακτήρα του θέματος των ιδίων πόρων και να προσπαθήσουμε να προσδώσουμε εδώ μια Ευρώπη, την εικόνα μιας Ευρώπης που κάνει μεταρρυθμίσεις, που μπορεί να επενδύσει, που αγαπά τους πολίτες, και δεν θα πρέπει μόνο να ζητάμε από τους πολίτες να αγαπούν τους, ε, την Ένωση, αλλά και η Ένωση να αποδείξει ότι αγαπά τους πολίτες της, τους νέους, τους ανέργους, τους πρόσφυγες, τη σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, να δείξουμε δηλαδή ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα δώσουν, θα παράγουν διαρκείς απαντήσεις. Ε, ένα ερώτημα και τελειώνω εδώ στα πλαίσια και της παρέμβασης την οποία έκανε η συνάδελφος Γουαρδιά Ζαμπάλε. σήμερα παίζετε εντός έδρας θα έλεγα, βρίσκεστε σε φιλικό περιβάλλον, είναι εύκολο εδώ, έχετε ένα ακροατήριο δεκτικό εν περιπτώσει, το έχουμε προετοιμαστεί σωστά, σας ακούσαμε, σας στηρίζουμε και θα δεχθούμε τις προτάσεις που θα κάνετε. Θα ήθελα όμως τα δικά σας ε, αισθήματα, όχι απέναντί μας, αλλά τα αισθήματα τα οποία νιώθετε εσείς όταν αντιπαρατήθεστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προθέσεις βλέπετε από πλευρά της Επιτροπής να υποστηρίξει ε, πραγματικά την χρήση της δυνατότητας της πρωτοβουλίας τους επόμενους μήνες και τι γίνεται στις συναντήσεις και στις αντιπαραθέσεις με το Συμβούλιο και πιθανώς και με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Θα ήθελα την κατάσταση αυτή να μας την περιγράψετε. Ε, Κυρία Νουριάντα. Δύο πατήσεις θέλω να κάνω. Καλημέρα σα. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερω σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε πρόταση η οποία ενδεχομένω να επιδεινώσει, να επιβαρύνει με πιο πολλού φόρου του πολιτέ μα. Γιατί ήδη υποφέρουν από τις πολιτικές λιτότητας από αυτά που συμβαίνουν με τις τράπεζες και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πιο πολλά. Έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να δώσουν και άλλα στην Ευρώπη όταν υπάρχει μεγάλη ενεργεία, όταν υπάρχουν ε, κρίση στο γαλακτοκομικό κλάδο. Ξέρω ότι υπήρξε παρέμβαση το περσινό έτος ύψους 500 εκατομμυρίων ε, και μίλησα με αγρότες από την δική μου επικράτεια που πήραν 500 ευρώ καθένας. Όλα αυτά όμως ε, καταλαβαίνετε ότι οξύνουν τον ευρωσκεπτικισμό ο οποίος ήδη υφίσταται και νομίζω ότι είναι δύσκολο να πουλήσουμε τις ιδέες αυτές στους πολίτες μας όταν βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν ε, ε, δουλεύει για αυτούς. Και φυσικά όλα αυτά ε, οξύνονται ιδιαίτερως από το Brexit. Το γεγονό λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα σε ό,τι αφορά την έλλειψη διαφάνειας, την έλλειψη της λογοδοσίας. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν όλα αυτά από τους πολίτες μας και να καταστούν διαφανή και κατανοητά. Εμείς μιλάμε, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τον προπολογισμό όσο έχει ήδη σε ό,τι αφορά και τους κανόνες για τους ίδιους πόρους και μήπως όλα αυτά δεν θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε και για μια, τι θα γίνει για μια σωστή κατανομή του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος. Προτού προχωρήσουμε και συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είχατε πει λοιπόν στην αρχή σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είστε υπεύθυνοι γι' αυτό, αλλά πρόκειται και για την ενοποίηση των ε, εθνικών οργανισμών και του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, σε ό,τι αφορά την συνάντηση δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σχόλια για την ε, ε, αξιολόγηση των πιστώσεων και των, ε, της πιστοποίησης των εθνικών και δημοσίων λογαριασμών προκειμένου να εναρμονιστούν και να τυποποιηθούν προκειμένου να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση των εγγράφων αυτών γιατί σήμερα πραγματικά είναι μεγάλη η πολυμορφία της. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο και τους υπόλοιπους ε, που άκουσαν πολύ προσεκτικά την παρουσίαση. Είναι πολύ σωστά τα σχόλια, πολύ εύστοχα τα σχόλια για την ενότητα και την ε, ε, ευκρίνεια του προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό και όπως είπατε θα πρέπει να προσέξουμε τη μέθοδο ώστε να έχουμε συγκρίσιμους εθνικούς με κοινοτικό προϋπολογισμό γιατί είναι πιο ε, καλύτερη η κατανόηση τους και των εθνικών αλλά και του ευρωπαϊκού. Είναι σημαντικό λοιπόν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να γίνει κατανοητός στους ευρωπαίους πολίτες και ένα από τα μηνύματα της ε, διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψης καλό θα ήταν να είναι ακριβώς αυτό. Περί και ευκρίνειας του κοινοτικού προπολογισμού. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Λαμασούρ που δεν είναι απλό μέλος της ομάδας ε, υψηλού επίπεδου, γιατί είναι και για την ομάδα αυτή, αλλά και για μένα προσωπικά ανεκτήμητη συνεισφορά με την ε, ευκρίνεια της σκέψης του και την πλούσια πείρα του. Είναι εξαιρετική η συμβολή του και η παρουσία του κυρίου Λαμασούρ αλλά και των υπόλοιπων εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομάδα υψηλού επίπεδου μας εξασφαλίζουν μία επικοινωνία σκέψης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ομάδας υψηλού επίπεδου, που είναι πολύ σημαντική. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια του κυρίου Λαμασούρ, γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και όντως οι συνέπειες του Brexit στη συζήτηση περί προϋπολογισμού θα μπορούσαν να είναι πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις του Brexit για τον προϋπολογισμό. Γιατί Brexit σημαίνει όχι ε, πια επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει και καμία άλλη επιστροφή πλέον. Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι εύλογο ένα τέτοιο επιχείρημα. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω In relation to είναι ένα κοινό στοιχείο όλων των ερωτημάτων. Πού βρισκόμαστε πολιτικά. Ποιο είναι το πολιτικό ύφος ή ο πολιτικός μας χώρος, η πολιτική μας θέση σχέση με τους ε, συνομιλητές μας που είναι τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Έχουμε ένα μόνο μέλημα και θεωρώ ότι η ομάδα μου συστήθηκε και εγώ ορίστηκα ως πρόεδρος αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου γιατί τα τρία θεσμικά όργανα ήθελαν να ακούσουν από εμά την αλήθεια. Γιατί Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να ακούγεται η αλήθεια, αλλά αν μη τι άλλο μια καλοπροαίρετη ε, στάση, η καλοπροαίρετη προσέγγιση της αλήθειας. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Και όσοι μου ανέθεσαν αυτά τα καθήκοντα, ε, θα είχαν επιγνώσει ότι και ε, όσο ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν δίστασα να χρησιμοποιήσω στο έπακρο τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άσχετα με τις αντιδράσεις των ε, κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων ε, της βιομηχανίας. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με την πλήρη χρήση των αρμοδιοτήτων, των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, των αρμοδιοτήτων γενικώ της Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί η Ένωση αυτή να ανταπεξέλθει στο έργο της και στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. και δεν είμαι πεπισμένος για την ε, ε, ωφέλεια της αυτομαστίγωσης που είναι μερικό, μερικές φορές κοινό χαρακτηριστικό όσων εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουμε ποια, ποιος είναι ο πολιτικός χώρος, η πολιτική μας θέση και θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω γιατί ξέρω ότι έχει κι άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ένα σύντομο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσος πολιτικός χώρος υπάρχει γύρω μας και τι πολιτικό περιθώριο έχουμε. Αλλά τίμα τη αποστολή μας ακριβώς είναι να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αυτό το πολιτικό χώρο, ώστε η διακοινοβουλευτική αυτή διάσκεψη δεν θα είναι μόνο να βρούμε πόσο πολιτικό χώρο έχουμε, ένα μικρός ή μεγάλος, αλλά και η διάσκεψη και η οριστική μας, η τελική μας έκθεση θα έχουν στόχο να αναγκάσουν τους αρμοδίους να σκεφτούν τις συνέπειες και ενδεχομένως να διευρύνουν και τον διαθέσιμο πολιτικό χώρο, το διαθέσιμο πολιτικό περιθώριο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να απαντήσω ενδελεχώς στις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Δεν φανταζόμουν ότι έφερα ελπίδα και αγαλίαση. Αυτό ξεπερνάει κάπως το στόχο μου. Πάντως χαίρομαι που έστω και κάποιες ε, πινελιές ε, συγκρατημένης εμπιστοσύνης έγιναν αντιληπτές. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Μόντι. Αυτά που είπατε θα μας επιτρέψουν να περάσουμε γαλήνιες διακοπές και να προετοιμαστούμε με επικοδομητικό τρόπο για την επιστροφή μας. Περιμένουμε λοιπόν το Big Bang στον δημοσιονομικό γαλαξία.